Okay, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήλθατε. Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε τώρα την συνεδρίαση της Επιτροπής μας για σήμερα. Στα δεξιά μου κάθεται ένας νέος συνάδελφος από την γραμματεία της Επιτροπής Σύντα, Όλιβερ. Ελπίζουμε να ξέρεις ε, τη δουλειά της Επιτροπής, αλλά νομίζω πως έτσι κι αλλιώς ε, ξέρει από σκληρή δουλειά και γι' αυτό θα θέλαμε να σε καλωσορίσουμε. Κυρία Χάουταλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μία επιστολή την οποία έστειλα σε εσάς και τους συναδέλφους την Παρασκευή. Όπως γνωρίζετε, στην ημερήσια διάταξη της 11 Δεκεμβρίου υπάρχει ακόμα ψηφοφορία για το ψήφισμα σχετικά με την ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βασίλειο του Μαρόκου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου για τη συμφωνία με την Μεσόγειο. Θεωρώ πως πρέπει να Σήμερα να, να δούμε τι θα κάνουμε. Πρώτον, υπάρχουν εγγυήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι η χνηλασιμότητα των προϊόντων ε, είναι εφικτή με τρόπο που να συμμορφώνεται προς το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έπειτα, κύριε Πρόεδρε, σέβομαι την αποφασή σα και την αποφασή των συντονιστών για να εξεταστεί εκεί το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων της ε, συναδέλφου Λαμών, αλλά να πω ότι για μένα προσωπικά η παρέτησή της από την ε, Ένωση EuroRenda είναι απόδειξη του ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν νομίζω πως ε, αυτό είναι σωστό και πως είναι κάτι που πρέπει να γίνεται στο Κοινοβούλιο ή έστω τουλάχιστον να μην ασχοληθεί αυτή η Επιτροπή με το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να εξετάσετε το αν επιτρέπετε να ψηφίσει στις 10 ε, Δεκεμβρίου. Εγώ νομίζω πως ακόμα όλα είναι ανοιχτά. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ε, σε ό,τι αφορά το Μαρόκο, να σας πω τα εξή Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μία σαφή διαδικασία για την ενίσχυση της συχνηλασιμότητας σχετικά με τα αγαθά που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε η Επιτροπή. Από όσο γνωρίζω, μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Έπειτα, σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, ε, κοίταξα με μεγάλη προσοχή τον εσωτερικό κανονισμό και αυτό είναι αρμοδιότητα του Προέδρου, ο οποίος και ενημερώθηκε, όπως ενημερώθηκε και ο επικεφαλής των ε, φιλελευθέρων, οι οποίοι είναι και οι δύο αρμόδιοι να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην έγκριση της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, τότε προτείνω να εγκριθεί με δύο τροποποιήσεις. Το σημείο 11, τα ζητήματα εσωτερικής αγοράς, να εξεταστεί μετά το σημείο 15. Έτσι λοιπόν, τα, τα σημεία 12 έως 15, δηλαδή η κοινή συζήτηση για τη Σιγκαπούρη, να ξεκινήσουν αμέσως μετά τις ψηφοφορίες. Υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν προτάσεις για αλλαγή. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 5ης Νοεμβρίου θα εγκριθούν λοιπόν εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σημείο 3. Αυτή η συνεδρίαση, όπως συνήθως, μεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο. Σας χαιρετώ όλους, λοιπόν, από το Ταλίνο στη Θεσσαλονίκη, από τη Λισαβόνα ως το Λούνεμπουργκ. Υπάρχει επίσης διερμηνία, γι' αυτό σας παρακαλώ να μιλάτε αργά, καθαρά και δυνατά, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να σας ακούσουν και οι διερμηνείς να μεταφράσουν αυτά που λέτε. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω κάποιους νέους συναδέλφους, ε, όπως ο ε, Όλιβερ Κρέντς που μόλις τον ε, καλωσόρισα. Και θα περάσουμε στο σημείο 4. Αποστολή της αντιπροσωπείας των ΟΣΑ στο Παρίσι της 21 Νοεμβρίου 2018. ΟΣΑ είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός στο πολυμερές ε, σύστημα εμπορικών συναλλαγών. Είναι μια δεξαμενή γνώσης και προβληματισμού σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την οικονομία. Και νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του ΩΣΑ σε αυτό το κλίμα προστατευτισμού που υπάρχει τελευταία. Η συνάντηση λοιπόν πήγε πάρα πολύ καλά. Συναντήσαμε πολλούς ε, εκπροσώπους του ΟΣΑ. Ήταν και ο πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρών και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την παρουσίαση των οικονομικών προπτικών για το 2019. Μάθαμε λοιπόν ε, πολλά σχετικά με αυτό και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ για την εμπορική πολιτική. Συμφωνήσαμε λοιπόν να υπάρχει στενότερη συνεργασία με τον ΟΣΑ στο μέλλον. Και η Τζουντ ήταν στην αντιπροσωπεία, οπότε θα της δώσω το λόγο γιατί θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ πολύ, Μπεν. Δεν περίμενα να πάρω το λόγο, αλλά Συμφωνώ μαζί σου, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η μερίδα. Αν καταλαβαίνω καλά, ήταν πρώτη φορά που υπήρχε μια επίσημη επίσκεψη της ε, ε, επιτροπής, της κοινής επιτροπής του Κοινοβουλίου στον ΩΣΑ. Ήταν λοιπόν ε, πλήρες το πρόγραμμα της ημερησίας διατάξης στο Παρίσι. Βρήκαμε ε, πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στις ε, συζητήσεις ανάμεσα στον ΟΣΑ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε τα ίδια περίπου θέματα και η βαρύτητα που δίνουμε σε αυτά είναι ε, παρόμοια. Υπήρξαν ορισμένα θέματα τα οποία νομίζω αξίζει να αναφέρουμε όταν ενημερώνουμε το κοινό για την Επιτροπή και καλό θα ήταν να το κάνουμε παρά το ότι υπάρχει το αρχείο κάπου στο διαδίκτυο. Λοιπόν, καταρχάς ε, οι πιστώσεις εξαγωγών. Στην Επιτροπή μας τους ερχόμενους μήνες θα συζητήσουμε τις συστάσεις της διαμεσολαβήτριας σχετικά με τις επιστώσεις εξαγωγών και νομίζω πως ε, μετά από τη συζήτηση αυτό που φάνηκε ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι κινητήριος δύναμη και προάγει τις ε, αξίες της, την διαφάνεια. Γι' αυτό νομίζω πως ε, φάνηκε στην ε, συζήτηση, φάνηκε επίσης και η σημασία της δέουσας επιμέλειας και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Με το Europax δημιουργείται μία, ένα, με ένα δυναμικό και πρέπει νομίζω, πως, πρέπει νομίζω να δράξουμε την ευκαιρία έτσι ώστε να διασφαλίσουμε μια πιο εξισορροπημένη εμπορική πολιτική στο μέλλον. Οι πιστώσεις λοιπόν εξαγωγών και ιδέουσα επιμέλεια είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία όπως και με τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συγκρούσεων. Και θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιμείνει στην τακτικότητα των μέτρων ελέγχου αυτής της δέουσας επιμέλειας. Σε συνεργασία φυσικά με τον Όσα. Δύο άλλα σημεία που θεωρώ εξίσου σημαντικά ήταν αυτή η μετάβαση, αυτή η αλλαγή άποψη των ΩΣΑ που παρατηρείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θεματολόγιο εμπόριο για όλους, για αυτήν την ε, αναδιάρθρωση της εμπορικής πολιτικής αυτό είναι και κάτι που απασχολεί πολύ την κοινή γνώμη και κατέστη σαφέ μετά από τις συζητήσεις ότι δεν πρέπει να βάζουμε νέα συσκευασία σε παλιές ιδέες, αλλά να δημιουργήσουμε νέα πολιτική που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών για τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και τις ανησυχίες επίσης των πολιτών για το πώς το εμπόριο επηρεάζει τις διάφορες περιφέρειες. Θεωρώ λοιπόν πως θα μπορούσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουμε έτσι γενικά το θέμα αυτό, να δούμε τι βγήκε από τις ε, συζητήσεις. Επίσης, από ό,τι φάνηκε δεν πρέπει να υπάρχει κατακαιρματισμός και αυτό βέβαια που είναι σημαντικό για μας είναι να δούμε πώς συνεργαζόμαστε με τις άλλες επιτροπές με... για το θέμα αυτό του Παγκόσμιου Θεματολογίου για το Εμπόριο. Αυτό όμως είναι εσωτερικό, είναι του Κοινοβουλίου περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι δύο μεγάλοι πυλώνες. Και ένα τελευταίο σχόλιο, επιτρέψτε μου, κάπως αρνητικό βέβαια. Με απογοήτευσε η συζήτηση για ένα συγκεκριμένο θέμα. όλες αυτές οι συγκρούσεις και εντάσει που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, το ντάμπινγκ, ο αθέμητος ανταγωνισμός, έχουν βρει πρόσφορο έδαφος στον τομέα της χαλιβουργίας και νομίζω πως ε, χρειάζεται να δούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πώς μπορούμε να θεσπίσουμε στιβαρά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση της ε, χαλιβουργίας. Αυτό φάνηκε νομίζω ότι η εργαλειοθήκη μας, όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ε, ανησυχίες του κλάδου, οι οποίες δεν είναι καινούριε, ε, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και θεωρώ λοιπόν πως ε, ως Επιτροπή θα μπορούσαμε να εξετάσουμε λίγο περισσότερο το τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και βεβαίως, ναι, η τελευταία συνάντηση για θέματα χάλιβα δεν ε, ε, μας προχώρησε και πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Μινέρ, ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Πρόεδρε. Η αποστολή όντως στον ΩΣΑ ήταν μια πολύ καλή αποστολή. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε βέβαια για όλα τα θέματα. Ήθελα να κάνω... Voor ongelimiteerde vrijhandel, maar handel gericht te reguleren. Ε, κοιτάξτε, πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να βρούμε κάποια στοιχεία για το εμπόριο, τα οποία να μας βρίσκουν όλους ε, ε σύμφωνους. Το θέμα της διατησίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν συζητήθηκε καθόλου από πλευρά του Κοινοβουλίου. Γιατί όμως... Ε, είναι γεγονός ότι ε, συζητήσαμε για κάποια θέματα, αλλά όχι τα ουσιαστικότερα και αυτά είναι ε, πολύ σημαντικά. Εν συμπεράσματι, όσα κάνει πολύ καλή δουλειά και χρήσιμη και ε, βεβαίως προσπαθεί στις πολυμερείς σχέσεις να ε, φέρει κάποιες λύσεις. Ωστόσο θα πρέπει να ε, φερθούμε πραγματικά, να συμπεριφερθούμε σαν να είμαστε βιομηχανοποιημένες χώρες και πραγματικά να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αφορούν και τον ανταγωνισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι, θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε στην ε, συνεργασία. Ε, το Φεβρουάριο ενδεχομένως ε, θα συμμετάσχουμε ως Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος, στο κοινοβουλευτικό δίκτυο του ο Σαχάιντι Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να ήμουν και εγώ εκεί, γιατί εκτιμώ ιδιαιτέρως αυτές τις κινήσεις, κυρίως δε αυτήν την ε, φιλοσοφική κατά κάποιο τρόπο εργασία την οποία ε, κάνει ο ΣΑ, προσπαθώντας να βρει όχι μόνο ε, στοιχεία και θεωρίες, αλλά και μεθοδολογία εφαρμογής αυτών των αρχών. Ε, ε, η υλοποίηση της, ε, του θεματολογίου του 2013 και οι βιώσιμες και τα, η στόχη τη βιώσιμη ανάπτυξη έγινε κάποια συγκεκριμένη συζήτηση γι' αυτό. Πρόεδρο, συζητήθηκε, αλλά όχι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πιο πολύ διασυνδέθηκε η συζήτηση με το ε, θέμα ε, της ανάγκης ύπραξης μιας συνεκτικής ε, στρατηγικής που θα καλύπτει όλους τους τομείς. Εκείνοι είπαν τι κάνουν εκείνοι από τη δική τους πλευρά και τι κάνουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς δεν ξέραμε και πολύ καλά τι να πούμε. Είπαμε ναι, ναι, υπάρχουν και διάφορες δομές. Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως είναι ένα σημαντικό θέμα και για μας. Πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε την εμπορική μας πολιτική ε, και οπωσδήποτε ε, για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει οπωσδήποτε να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Ίσως Φεβρουάριο του 2019 λοιπόν έλεγα, ε, ίσως συμμετάσχουμε στην συνάντηση του κοινοβουλευτικού δικτύου όσα, έτσι ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η σχέση μας. Επόμενο σημείο είναι το σημείο 5 το οποίο αφορά την κατάσταση των συνεχισμένων διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. Ε, πρώτα απ' όλα για το θέμα της ρήτρα διασφάλισης, ο κύριος Χάνσεν εξ του Κρίστοφερ Φιέλνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κύριου Φιέλνερ ο οποίος ε, δυστυχώς λόγω απρόβλεπτων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Διαβάζω λοιπόν αυτά που μου άφησε. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή γιατί δούλεψε πάρα πολύ καλά ε, και... Α, όχι, αυτό είναι το επόμενο θέμα. Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Α, δεν, μόνο αυτό μου έχει δώσει όμως. Τώρα συζητάμε για τον τριμερή διάλογο για, την οριζόντια, ε, για την κανονισμό για την οριζόντια ρήτρα διασφάλισης. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο κατάφερε να περάσει πολλές από τις ε, τροπολογίες όσον αφορά ε, τον έλεγχο των κεφαλαίων TST, τις δυνατότητες για τα συνδικάτα να διερευνήσουν καταστάσεις, δυνατότητα εστίασης επίσης σε πιο ευαίσθητα προϊόντα, και επίσης δυνατότητα να μελετηθούν τα προβλήματα των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Η συζήτηση αυτή έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι ε, ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί έχουμε άλλωστε και στην δική μας ημερήσια διάταξη εμπορικές συμφωνίες και επομένως αυτό το θέμα της οριζόντιας ρήτρας διασφάλισης είναι κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Ο κύριος Φιέλνερ δούλεψε πάρα πολύ καλά και το αντιμετώπισε σωστά. Βεβαίως θα έχουμε σύντομα και επόμενο τριμερή διάλογο για το θέμα των ποσοστώσεων στο ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου Έχουμε ε, αύριο τριμερή διάλογο για αυτό το θέμα και ίσως, δεν το ξέρουμε βέβαια, κανείς δεν ξέρει, ίσως προκύψει πρόοδος και φτάσουμε κοντά στο, στην τελική ευθεία. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε και ένα τρίτο νομοθέτημα υπό Αυστριακή ε, ε Προεδρία. Και ίσως λοιπόν μπορέσουμε να κλείσουμε αυτά, αυτούς τους φακέλους. Θα υπάρξει βέβαια κι άλλος ένας ανοιχτός φάκελος ε, που είναι ο έλεγχος εξαγωγών. Προχωράμε. Το Συμβούλιο ενδεχομένως ε, εντός του Δεκεμβρίου θα εγκρίνει την εντολή ε, της διαπραγμάτευσης και θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις εντός του Δεκεμβρίου. Ευελπιστούμε δε ότι θα υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωση των διαδικασιών ε, εντός της τωρινής θητείας και τότε το Κοινοβούλιο ε, θα δείξει για μία ακόμα φορά ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικό ε, και έχει άσους κρυμμένους στο μανίκι. Πολλές δυνατότητες έχει το Κοινοβούλιο. Προχωράμε λοιπόν το θέμα της εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών Δυστυχώς ε, δεν ξέρω πού βρισκόμαστε, ε, πόσο έχουν προχωρήσει αυτές οι συζητήσεις. Ε, δεν είναι εδώ και η κυρία Μόσκα, θα τα πούμε αργότερα. Σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως αφορά την εφαρμογή του κανονισμού σίγμα γάμα πι. Κύριε Χάνη, σας ξαναδίνω το λόγο. Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Ο κύριος Φιόλνερ λοιπόν μου ζήτησε να διαβάσω το εξή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πολύ καλή δουλειά που αποδεικνύει ότι ε, ε, ε, μπορούμε να επιτύχουμε και τη μείωση της φτώχειας και την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης και την κάλυψη των οικονομικών συμφερόντων μέσω αυτής της νέας συμφωνίας. Αναφερόμαστε στο σήμα ΓΑΜΑΠΗ ε, των Ηνωμένων ε, Εθνών και σημειώνουμε δύο μεγάλες διαφορές τις οποίες ε, υποστηρίζει ο εισηγητής. Μεγαλύτερη αστίαση όσον αφορά την διασύνδεση των γενικευμένων προτιμήσεων με τις ε, με τους βιώσιμους στόχους ε, ανάπτυξης. Βεβαίως μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις ε, εάν η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συντονιστούν καλύτερα με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις της, καθώς επίσης και με τις εν λόγω χώρες θα πρέπει να προσέξουμε την, ε, το θέμα της διαφοροποίησης. Ε, αυτή η ε, δυνατότητα να φτάνουμε στον πραγματικό δικαιούχο είναι ένα σημείο το οποίο μας προβληματίζει. Πιστεύουμε ότι όλο και περισσότερες χώρες θα πρέπει να συμπαραταχθούν σε αυτή τη διαδικασία. Aid for Trade, περισσότερες χώρες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτήν την διαδικασία. Θα πρέπει οπωσδήποτε και οι υπηρεσίες να συμπεριληφθούν ε, σε αυτήν την διαδικασία. Το Κοινοβούλιο έχει δουλέψει πάνω στο θέμα αυτό μέσω ψηφισμάτων και πρέπει να προχωρήσουμε τώρα ε, θα πρέπει οπωσδήποτε και ο περιβαλλοντικό αντίκτυπο να μελετηθεί υπεραιτέρω και χρειαζόμαστε συγκεκριμένε δράσει, έτσι ώστε ε, στον επόμενο κανονισμό αυτό να γίνει σαφέ. Ο εισηγητή γνωρίζει ότι υπάρχουν τροπολογίε, αλλά υπενθυμίζει στου συναδέλφου ότι εδώ στόχο είναι η mid-term review. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο ε, θα έχουν οι σκιώδεις εισηγητές, ε, η κυρία Μόσκα. Α, την εκπροσωπή συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δυστυχώς δεν είναι εδώ η συντονιστριά μας, γι' αυτό παίρνω εγώ το λόγο εξ ονόματός της. Αγαπητέ εισηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, ιδιαίτερε ευχαριστίες στον ε, εισηγητή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για το χρονοδιάγραμμα που έχει υποβάλει. Η έκθεση έφτασε με ε, καθυστέρηση. Ε, επιμένω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει σχετική γνωμοδότηση. Το θέμα των γενικευμένων προτιμήσεων είναι ένα σύστημα που μπορεί πραγματικά να υποστηρίξει την ανάπτυξη η βιωσιμότητα μεταξύ άλλων βασίζεται και σε την ε, ε, αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, πράγμα στο οποίο αντιτίθονται βεβαίως οποιασδήποτε καθυστερήσεις. Η ενίσχυση της ε, συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών μόνο και η ενισχυμένη επιτήρηση μπορούν να βελτιώσουν τις, την κατάσταση. Κατά την έννοια αυτή έχω υποβάλει τροπολογίες. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, χώρες ε, να δέχονται την βοήθεια αυτή και να την χρησιμοποιούν χωρίς στόχο σωστό. Θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να ελέγχεται διαρκώς η αποτελεσματικότητα της χρήσης. Όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών, προτείνω να συμπεριληφθεί στην ε, έκθεση ένας ε, ε, σαφής μηχανισμός προσφυγών και υποβολής καταγγελιών. Κατά την έννοια αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε και η Κομισιόν να είναι ιδιαίτερα αποφασιστική όταν συζητά την συμμόρφωση των χωρών αυτών ε, με τις ε, αρχές της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας καθώς επίσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί παρά μόνο με τον έλεγχο ότι ε, οι χώρες ε, είναι σύμφωνες και σέβονται τις αρχές που έχει θεσπίσει η Κομισιόν. Από, σε όλες τις χώρες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε γιατί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντί να βελτιώνεται βαίνει επιταχύρω. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Και η κατάσταση σε σχέση με τους πολίτες των ΗΠΑ και τους πολίτες της Ευρώπης, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που ζουν στις χώρες αυτές θα πρέπει ιδιαίτερως να προσεχθεί. Τα προγράμματα ε, ε, ε, τα προγράμματα των γενικευμένων προτιμήσεων, εάν δεν ελεγχθούν σωστά, μπορούν να στραφούν εναντίον του θεμητού ανταγωνισμού και να οδηγήσουν σε dumping. Θα πρέπει οπωσδήποτε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Κομισιόν, η Κομισιόν δηλαδή να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα και στους πολίτες ε, των χωρών και στις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω δύο βασικά πράγματα, αλλά Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κρίστοφερ για την ε, δουλειά που έκανε. Δεν είναι εδώ, αλλά θα μεταφερθούν τα λόγια μας ε, και θα προχωρήσουμε με τροπολογίες. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που βλέπω ότι ο Κρίστοφερ δεν προχώρησε αναχώρα, αλλά επέλεξε να προσεγγίσει συνολικά το σύστημα των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Τα δύο πράγματα που ήθελα να πω. Το πρώτο αφορά τη διαφοροποίηση. Χαίρομαι που ο Κρίστοφερ υπογράμμισε αυτό το θέμα στην έκθεσή του. Πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να τύχει της προσοχής μας. Γιατί δεν έχουμε επιτύχει ακόμα ε, τα αποτελέσματα που θέλαμε να δούμε σε ό,τι αφορά τις ε, εξαγωγές των χωρών. Οι χώρες έχουν τη τάση να ε, εστιάζουν στις, ε, στα δυνατά τους σημεία, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερες ό,τι αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ενδεχομένως να δρομολογήσουμε κάποια προγράμματα. Το GSP Plus το ειδικό καθεστώς επιτρέπει σε κάποιες χώρες να εξάγουν ε, προϊόντα σε εμά. Έχουν όμως ως αποτέλεσμα να αυξάνουν και τις ε, εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτές τις ε, χώρες. Άρα θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά σε αυτό το τομέα. Τέλος, το θέμα που ανέφερε και η συνάδελφος υπάρχουν ελλείψεις που αντιβαίνουν στους στόχους μας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να επιδείξουμε περισσότερη φαντασία. Δεν είναι όλα μαύρα ή άσπρα. Σήμερα έχουμε ένα ε, γενικό καθεστώς και αύριο δεν υπάρχει. Πρέπει να δούμε ποιες μπορεί να είναι διαφορετικές ε, προσεγγίσεις. Το ανέφερε αυτό το θέμα ο Κρίστοφερ στην έκθεση, όταν μιλάει για πιο στοχευμένη προσέγγιση ε, και περιορισμό σε συγκεκριμένους τομείς, σε παραβιάσεις τα πιστοποιητικά εξαγωγών από συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Νομίζω ότι εδώ έχουμε κάποιες βάσεις προκειμένου να προχωρήσουμε παραπέρα και να φροντίσουμε να προτρέψουμε τις αρνητικές ε, συνέπειες προς τις χώρες τις οποίες θέλουμε να προστατεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λελόν δεν είναι εδώ. Η κυρία, η κυρία Ρης. πράσινη και η γκουε είναι ίση, άρα ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Το κανονισμός ε, ε γάμα σίγμα π είναι πολύ σημαντικό μέσο. Λάβαμε το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Φίλντερ. Δεν προσθέτει βέβαια πολλά στοιχεία στην έκθεση της ε, Επιτροπής. Φαίνεται πως η μόνη αλλαγή που έχει η Κομισιόν στο μυαλό της για τη χρήση αυτού του μηχανισμού δασμολογικών προτιμήσεων είναι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Η Κομισιόν όμως θα, καλό θα ήταν να μας πει πώς βλέπει τα πράγματα, πώς θα μπορούσε να συμμετέχουν οι ε, οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών. Ε, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η δημοκρατία σε χώρες που, όπου στην πραγματικότητα η δημοκρατία δεν λειτουργεί πολύ καλά. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι το εξής. Μπορούμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις χώρες που υπάγονται, για παράδειγμα, στο ειδικό καθεστώς. Πρέπει ε, αυτός ο στόχος είναι να ε, βοηθηθούν αυτές οι χώρες να, είναι, να δεσμεύονται προς την επίτευξη συγκεκριμένων ε, στόχων. Χρειάζεται μία προοδευτική εφαρμογή των προτιμήσεων θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως ένας ε, μοχλός. Αυτό αφορά συγκεκριμένα το Μιανμάρ και την Καμπότζη. Το βασικό ερώτημα είναι ε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Ε, επίσης, το θέμα των αποκλειστικών ζωνών παραγωγής. Η ομάδα μου πιστεύει ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το θέμα όταν μιλάμε για την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων οι αποκλειστικές ζώνες παραγωγής ε, γίνονται όλο και πιο σημαντικές σε ό,τι αφορά τις γενικευμένες ε, προτιμήσεις, αλλά συνήθως αποκλείονται από τις διεθνείς συμβάσεις. Η Κομισιόν θα ήταν έτοιμη να συζητήσει αυτό το θέμα. Και σε ό,τι αφορά ε, όλα εκτός από όπλα, ε, πρέπει να τύχει και αυτό το θέμα της προσοχής μας. Ε, γιατί να μην, για να, τι να μην δίνονται κίνητρα ε, για, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία όλων. Τέλος, πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να συμμετέχει στους ελέγχους για τον καθορισμό των δικτών. Και τελευταία ε, παρατήρηση, το Μπαγκλαντές και η βιώσιμη ανάπτυξη ε, έχουν προχωρήσει πολύ ε, σε αυτό το θέμα. Στην αρχή η Επίτροπος Μάνστρομ είχε πει ότι αυτό το σύμφωνο θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες, το Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μπορούμε αυτό να το λόβουμε υπόψη Μπορούμε να λάβουμε υπόψη μα αυτού του στόχου του Συμφώνου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη περίπτωση Μπαγκλαντέ. Η Ανμαρή Μινέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σήμερα μιλάνε κυρίως οι αντικαταστάτες. Ε, μιλήσω κι εγώ εξ ονόματος ε, μιας συναδέλφους. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών, των, της χρηστής διακυβέρνησης. Χαιρετίζουμε την διάμεση αξιολόγηση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις γενικευμένες προτιμήσεις και καλασορίζουμε το ε, γεγονός ε, ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές ε, των χωρών που υπάγονται στο καθεστώς όλεκτος εκτός από όπλα. Η αξιολόγηση συμμετέχει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Χαιρετίζουμε και το, το ότι υπογραμμίζεται η σημασία της διαφάνειας. Ε, και σημαντική είναι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ε, του ιδιωτικού τομέα. Υπενθυμίζουμε ότι για να ενισχυθεί η διαφάνεια, ο έλεγχος και η υπαγωγή στο καθεστώς GSP Plus πρέπει να είναι προσβάσιμος. Ε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που δίνονται από ε, τρίτους ε, με στόχο την ε, εφαρμογή των διεθνών συμβόσεων. Η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη τι απειλέ ε, προς τα συνδικάτα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμμετοχή της κοινωνίας των ε, πολιτών και τη δρομολόγηση διαλόγου, Μια και σημασία είναι, ε, εν τέλει, έχει, σημασία εν έχει η συμμόρφωση με τις νομικές ε, διατάξεις. Ενθαρρύνουμε λοιπόν την Κομισιόν να επεκτείνει το καθεστώς όλο εκτός από όπλα και σε άλλες ε, χώρες. Η Κομισιόν πρέπει να θέσει συγκεκριμένους δίτες, συγκεκριμένους στόχους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και να ε, λάβει υπόψη τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εφαρμογή της εμπορικής ε, πολιτικής. Πρέπει να προβλεφτεί μηχανισμός προσφυγών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπλέον, η μείωση των ε, δασμών πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχους. Οι τροπολογίες μας θα εστιάσουν σε αυτά τα θέματα και ο εισηγητής θα το λάβει υπόψη του. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια λοιπόν. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βάλτερ Χατούμ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω όμως και εγώ μια ερώτηση πριν από αυτό. Αυτή τη στιγμή συζητείτε το ενδεχόμενο να πάρουμε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων από την Μιανμάρ. Εσείς θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε πώς θα γίνει όλη η διαδικασία. και ποιοι είναι οι, διάφοροι, οι διάφορες ενδείξεις που έχετε για την έκφαση της ε, συζήτησης για το ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους πολίτες της Μιανμάρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής ΙΝΤΑ, καθώς και την ε, αξιολόγηση. Πρόσφατα έγινε συζήτηση στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, και είδα ότι συζητήθηκαν παρόμοια θέματα με αυτά που εξετάζετε εσείς. Και κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας ότι είναι πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί ως συνομοθέτη στον κανονισμό για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Νομίζω πως έχετε πάει πάρα πολύ καλά και πως ε, έτσι κι αλλιώς ο κανονισμός από μόνος του είναι ένας πολύ καλός ε, κανονισμός. Επίσης, εκτιμούμε την έμφαση που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ω μέσο για την ανάπτυξη, το οποίο φαίνεται και από τις συστάσεις σας. Νομίζω πως είναι μία ε, σαφέστατη ε, δήλωση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το θεματολόγιο της για το εμπόριο, ιδιαίτερα σε σχέση με άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με ορισμένα από τα συμπεράσματα, δηλαδή ότι το σύστημα αυτό ωφελεί τις φτωχότερες χώρες, ότι οι δικαιούχοι για το όλα εκτός από όπλα ανέβηκαν κατά 62% και ότι σε άλλους τομείς ανέβηκαν επίσης, κατά 54%. Επίσης, οι ρυθμοί προσαρμογής είναι ενδεικτική του ωφέλους που έχει το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για τις χώρες αυτές. Και κάτι άλλο, να πω ότι όλα αυτά δεν έγιναν εις βάρος της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω εδώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, αλλά και ότι οι δικαιούχοι στις τρίτες χώρες ε, μειώθηκαν από το 6% στο 4%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της έκθεσης, από ό,τι φαίνεται υπάρχει αντίκτυπος και στους ε, πολίτες και στα εργασιακά και στο περιβάλλον. Είναι ωστόσο αρκετά δύσκολο να γίνει ε, λεπτομερής αξιολόγηση. Ε, βέβαια, θα επανέλθω στη Μιανμάρ, να σας πω, δεν το ξεχνώ, αλλά το θέμα με τα εργασιακά δικαιώματα στο Πακιστάν είναι ένα θέμα που παραμένει. Η κατάσταση με τη διαδικασία εξαγωγών είναι κάτι που συζητήσαμε και να σας πω ότι ο, η νέα κυβέρνηση έχει και ένα νέο γενικό εισαγγελέα στο Πακιστάν, ο οποίος στο σύνταγμα του Πακιστάν ε, απαγορεύεται η κακή μεταχείριση των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν ε, υπήρχαν δεσμεύσει από πλευρά κυβέρνηση του Πακιστάν για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Τώρα σε ό,τι αφορά τι ε, Φιλιππίνες, η κυβέρνηση είναι θετικά προσκύμενη στην εφαρμογή του ε, GSP-SYN. Σε ό,τι αφορά την θανατική ποινή πέρασε ένα νόμο για την κατάργηση τη στο Κογκρέσο και χάρη στην Επίτροπο Μάλμστρομ αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η επανεισαγωγή τη θανατική ποινή δεν έγινε πραγματικότητα. Και συνεργαζόμαστε βεβαίως με τις κυβερνήσεις για αρκετά θέματα. Τώρα, ε, οι συστάσεις που αναφέρατε ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Έχω να πω κάτι σχετικά με την διαφάνεια όμως. Ε, σίγουρα μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα υπό τον υφιστάμενο κανονισμό, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τον επόμενο και εξετάζουμε το πώς θα γίνει αυτό. Τώρα, ε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, γίνονται συναντήσεις ε, ε, και πριν μεταβούμε στις χώρες αυτές, αλλά και επιτόπου. Και σίγουρα η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έπειτα, συνεργασία και εταιρική σχέση με τους δικαιούχους. Χρειάζεται να ενισχυθεί έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού για το πώς ε, να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και όλο το σκεπτικό πίσω από αυτό το σύστημα είναι να προσελκύσει νέες επενδύσεις σε τομείς οι οποίοι ε, υστερούν μέχρι τώρα. Αυτό θα ωφελήσει και την βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο έλεγχος τώρα ε, είναι πλήρης. Υπάρχουν 27 συμβάσεις και εμείς προσπαθούμε αντί να γίνει μια γενικότερη, ευρύτερη συζήτηση να κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες, να δούμε ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε όπως κάναμε και στο Πακιστάν ε, και ζητήσαμε από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα μέχρι τον επόμενο Ιούνιο για τις ε, λήψεις ε, που έχουν εντοπιστεί αλλά στην έκθεση υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρήση του συστήματος και η Επίτροπος ε, Μάλμστρομ έχει αναφερθεί ε, στον ενισχυμένο έλεγχο της συμφωνίας σε τα πάντα εκτός από όπλα. Στην περίπτωση της Μιανμάρ και της ε, Καμπότζης θα γίνει και εξακολουθικός έλεγχος. Στις αρχές του 2017, στην ανακοίνωσή μας ε, εξάλλου, αναφερόμαστε ε, στην αξία του GSP Plus και στα διδάγματα που θα πρέπει να αντλήσουμε έτσι ώστε στο μέλλον να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τέτοιες περιπτώσεις ε, κυρίως που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα, όχι τόσο το περιβάλλον. Νομίζω πως η δύναμη ε, του πακέτου της ε, Επιτρόπου Μάλιμστρομ θα έχει μεγάλο αντίκτυπο όχι, όχι μόνο στην Καμπότζη και στη Μιανμάρα αλλά και στο στάδιο της αξιολόγησης σε άλλες χώρες οι οποίες δεν ε, χρησιμοποιούν το μηχανισμό απόσυρσης. Όταν πήγαμε στο Πακιστάν, λίγο μετά την παρουσίαση της δέσμης μέτρων της Επιτρόπου Μάλιμστρομ, είδαμε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ενασχόληση με το σύστημα αυτό και προσπαθούμε να διευρύνουμε τις καλές αυτές πρακτικές και αλλού. Τώρα, σε ό,τι αφορά του ε, ελέγχου τη αξιολογή τη βιομηχανία, νομίζω πω πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία. Γι' αυτό και μα ικανοποιεί πάρα πολύ το έργο τη Επιτροπή Ανάπτυξη, διότι στέκεται ακριβώ αυτό στου κανόνε προέλευση, ε, σε τελωνιακά ζητήματα, σε δασμού. Γι' αυτό λοιπόν ε, συνεργαζόμαστε στενά με αυτήν την Επιτροπή. Αυτοί είναι οι τομεί στους οποίους ε, θεωρούμε ότι μπορούμε ήδη να ξεκινήσουμε δουλειά. Στο πλαίσιο του επόμενου κανονισμού, βέβαια, θα εξεταστούν άλλα ζητήματα τα οποία είναι δύσκολο να επιληθούν αμέσως. Όμως είναι καλό να τα κοιτάζουμε εγκαίρως, έτσι ώστε μέχρι του χρόνου να έχουμε οδηγηθεί σε κάποια συμπεράσματα. Ε, για κάποια ζητήματα που υπάγονται αυτή τη στιγμή στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, αλλά για παράδειγμα πώς να ενισχυθεί ο θετικός αντίκτυπος για το περιβάλλον, πώς να συμπεριληφθούν περισσότερες συμβάσεις στο σύστημα, πώς ε, να μειωθεί ο αριθμός των ε, περιπτώσεων απόσυρσης το σημείο για τη συσσόρευση κανόνων προέλευσης ε, εξετάζεται υπό τον υφιστάμενο κανονισμό. Χρησιμοποιείται στην περίπτωση Καμπότζης και της Μαλαισίας, όμως πρέπει να ζητήσουμε να εφαρμοστεί. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε από κοινού τις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και συμπερασματικά Καλωσορίζουμε την έκθεση της Επιτροπής ΙΝΤΑ αλλά και την ενδιάμεση αξιολόγηση. Θα ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε αμέσως ορισμένα από τα ευρήματα της έκθεσής σας. Ε, ωστόσο, νομίζω πως πρέπει να υποφεληθούμε από το ότι ε, μπορούμε να συνδυάσουμε και το εμπόριο αλλά και το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Ο νέος κανονισμός ελπίζω να είναι τόσο ενδιαφέρον για την Επιτροπή σας όσο και ο προηγούμενος, διότι θα τεθεί σε ισχύ από το 2024, όμως χρειάζεται πριν την ε, ημερομηνία αυτή να γίνει μεγάλη προεργασία. Αυτά λοιπόν από μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα έχω να προσθέσω σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση και τις προοπτικές. Η Επιτροπή ε, αυτή τη στιγμή εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπιση συγκεκριμένων προτιμήσεων για προϊόντα τα οποία θα ε, πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όχι δηλαδή να καλύπτεται μια ολόκληρη χώρα, αλλά ένα συγκεκριμένο είδος, ένα συγκεκριμένο τύπος παραγωγής. Και επανέρχομαι στη μια για το, τη δεύτερη ερώτηση. Θεωρείτε πως αυτό το blog, αυτό το σύνολο είναι το κατάλληλο μέσο για να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση των ε, τρίτων χωρών. Ε, δεν είμαι πεπισμένος ότι ούτε, ε, ούτε τα blog, ούτε... Τα blog, ούτε το Twitter είναι τα κατάλληλα μέσα για να προχωρήσουμε και για να επικοινωνήσουμε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι στην περίπτωση της Μιανμάρ θα πρέπει να γίνει επίσημη έρευνα Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά ε, την πρώτη σας ερώτηση, ενδιαφέρουσα ερώτηση, αυτή, αυτό δεν είναι δυνατό όμως υπό τον παρόντα κανονισμό. Όμως, όταν ήμουν στις ε, Φιλιππίνες, είδα ότι δουλεύουμε πάνω σε έναν κανονισμό. Ας πούμε, αυτές που οι εταιρείε οι οποίες δουλεύουν ε, στο, στην ένδυση μπορεί να μην έχουν άδεια εξαγωγών. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτές, ε, ε, πρόκειται, αυτές είναι ε, πρωτοβουλίες συγκεκριμένων χωρών. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να διευκολύνουμε το εμπόριο γενικότερα, άρα προσεκτικά και τα κριτήρια. Όσον αφορά την Μιανμάρ, ξέχασα να απαντήσω στην ερώτησή σας που αφορά ποιες, το, το θα είναι οι επιπτώσεις για τον κόσμο εκεί η Κομισιόν. Συζήτησε το θέμα αυτό τον προηγούμενο μήνα στην συνάντηση υψηλού επίπεδου. Είναι 500.000 οι εργαζόμενοι περίπου στον τομέα της ένδυσης, κυρίως νέες ε, γυναίκες οι οποίες ε, στέλνουν και χρήματα για να υποστηριχθεί η γεωργία στα χωριά τους και αυτά και επομένως ε, εάν σταματήσει η διαδικασία αυτή τότε θα γίνει πολύ ευάλωτος αυτός ο πληθυσμός όσον αφορά την αξιολόγηση, ναι, εάν δεν χρησιμοποιήσει κανείς τον withdrawal mechanism, τον μηχανισμό απόσυρσης, ίσως χάσει κανείς την αξιοπιστία του. Τώρα, πώς γίνεται η πληροφόρηση και η επικοινωνία, να σας πω ότι το σημαντικό είναι ο αντίκτυπος όσον αφορά τις διαδικασίες. Ε, ε, ε βεβαίως υπάρχει συγκεκριμένες δυνατότητες αναφέρονται στον κανονισμό ε, για τις γενικευμένες ε, προτιμήσεις, ε, δηλαδή γίνονται αξιολογήσεις τους έξι μήνες, μετά στους ξανά άλλους έξι μήνες και γίνεται μετά η τελική αξιολόγηση και η χώρα έχει κάποιες εβδομάδες για να απαντήσει. Ναι, είναι λίγο χρονοβόρα η διαδικασία, αλλά επιτρέπει ταυτόχρονα και διάλογο με τους εμπλεκόμενους και εδώ και στην τρίτη χώρα. Το κύριο μήνυμα λοιπόν είναι ότι εάν ε, πρέπει να ξεκινήσει ε, ε, κάποια αξιολόγηση η οποία θα οδηγήσει σε πρόσκαιρη απόσυρση, θα πρέπει να σκέφτεστε μόνο εν τέλει το, το βαθμό πίεσης και τη δυνατότητα πίεσης που έχουμε. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να έχουμε εμείς κοινή θέση. Τώρα το blog ε, δεν είναι η μόνη δυνατότητα επικοινωνίας, είναι ένας από τους τρόπους. Απ' την άλλη πλευρά να πω ότι ε, κάτι που δεν ήταν δεδομένο συνέβη, δηλαδή άνοιξε τις πόρτες της η για την αποστολή ε, και ήταν αρκετά υψηλό το επίπεδο επικοινωνίας, έτσι ώστε ενδεχομένως να έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Πρόεδρος, ωραία. Επομένως θα ξεκινήσει η αξιολόγηση για τη Μιανμάρα. Όχι, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, λέει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ε, θα δούμε αν ναι ή όχι θα γίνει μια ε, αξιολόγηση ε, και εάν θα ξεκινήσει η διαδικασία αν θα ξεκινησει η διαδικασια συμβουλιου και η συμβουλευτική συγγνώμη διαδικασία και θα δούμε, θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία. Πρόεδρος, εκτός μικροφώνου οι διερμηνείς δεν ακούν. Νομίζω ότι τα είπατε τόσο διπλωματικά, είσαστε έτοιμος για να γίνετε διπλωμάτης. Ε, κύριε Χάνης, παρακαλώ για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Μια και απλώς αντιπροσωπεύω τον κύριο Φιόλνερ, εγώ ε, να πω ότι σημείωσα προσεκτικά τα όσα είπατε, θα τα διαβιβάσω στον κύριο Φιόλνερ ε, και εξ ονόματός του σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. 19 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι λίγη προθεσμία υποβολής τροπολογιών, ακριβώς το μεσημέρι. Perfect. Ωραία. Φτάνουμε τώρα ε, στις ε, ψηφοφορίες. Ε, μάλλον όχι, πρέπει να διακόψουμε για πέντε λεπτάκια όμως. Ε. Ναι. Okay, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτο θέμα είναι το 7 της ημερησίας διατάξεως. Πριν όμως θα κάνουμε μία δοκιμή ψηφοφορίας, άρχεται η ψηφοφορία. Ελέγχουμε τώρα. Has everybody voted? Ψήφισαν όλοι. So this Mr. Martin is the last one here. Κύριε Μάρτιν, ψηφίστε κι εσείς. Ωραία. Έγινε και ο έλεγχος. Όλα είναι καλά. Fine. And we start now with, uh, item seven. Προχωράμε λοιπόν εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κολομβία και το Περού. Ο κύριος Φίσας είναι ο εισηγητής. Ε, τροπολογία 13, παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχέσε εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχέσε απορρίπτεται. 29 υπέρ. Against, abstention rejected. 30 in favor. Against, abstention adopted. 31 in favor. Against, abstention rejected. 32 in favor. Against, abstention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 Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται συμβιβαστική έξι νέο υπέρ κατά αποχέσε εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ ναι, είναι η παλιά προφορική. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η 50, Χάιντι Χαουτάλα, έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ η τροπολογία 50, το δεύτερο τμήμα, να ψηφιστεί ως προσθήκη ε, της συμβιβαστικής 7 που μόλις εγκρίναμε. Να ζητήσουμε από την Κομισιόν ε, να μας δώσει και ε, συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τις γυναίκες, τους αναπήρους κλπ. Και μέσα στα εξαγωγικά της στοιχεία. Πολύ ωραία το δεύτερο τμήμα της 50 ως προσθήκη στην συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 52 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Δεν είμαι σίγουρος, λέει ο Πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 73 ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 νέο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, ε, συγγνώμη, συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές Καλύτερα να κάνουμε μία επαλήθευση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας και απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία επί της τροποποιημένης ε, εκθέσεως με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Ω, με μεγάλη πλειοψηφία ευχαριστούμε πολύ κύριε Φίσα και συγχαρητήρια. So, next point is... Επόμενο σημείο, 8, έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνία Σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική. Ο κύριος Μπέγκε είναι ο εισηγητή. Και ξεκινάμε με την τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται συμβιβαστική 5 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική υπαλλήθευση επί της τροπολογίας 41 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απερίφθη τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 56 με προφορική τροπολογία. Στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά προτιμώ να το ελέγξουμε. Ε, ψηφίζουμε λοιπόν 56 με προφορική τροπολογία στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας. Άρχεται η ψηφοφορία πέρασε και εγκρίνεται. Τροπολογία 51 δεύτερο τμήμα. Αυτό καταπίπτει γιατί έχει εγκριθεί το δεύτερο τμήμα της 56. Ε, τροπολογία 54 δεύτερο τμήμα. Και αυτό καταπίπτει. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι και σίγουρος. Ελέγχουμε την τροπολογία 58. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται πέρας. Και α, δεν έγινε δεκτή. 59 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Ψηφίζουμε στο πρώτο, για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος αν έχει απορριφθεί καλύτερα να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας και έχει απορριφθεί όντως Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά, αποχές. Καλύτερα να επαληθεύσουμε επί της ε, τροπολογίας 23 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται.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 Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία πάντα με ηλεκτρονικό τρόπο. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας και μπράβο και συγχαρητήρια γιατί ενεκρίθη με μεγάλη πλειοψηφία. 27 ψηφί υπέρ, μία κατά. Point nine. Σημείο 9. Θέσπιση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας. Ο κύριος Μπορέλη ήταν συντάκτης. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Ψηφοφορία επί της 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε. Επί τις 12. Ε, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας, ελέγξουμε. Ας ψηφίσουμε. Άρκετη ψηφορία. ψηφοφορία. Επί της 18. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ε, ας ψηφίσουμε επί της 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23, 23 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, ε, επί, ψηφοφορία από 28, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία Πέρες εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία επί της 50. Πέρας. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ελέγχο, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και για το σύνολο της έκθεσης, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συγχαρητήρια, κύριε Μπορέλη. ότι τώρα θα περάσουμε στο ένα από τα πιο σεξι κομμάτια. Το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα. Συμβαστική 10, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Έλεγχος. φορεί επί της 105. Πέρας. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Έλεγχος. Ψηφορία επί της 106. Πέρας. Απορρίπτεται. 107 D υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφοφορία επί της ε, συμβαστικής 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 108D. Όχι, καταπίπτει. 114 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, ψηφοφορία, ε, ψηφορία επί της 114, πέρας, απορρίπτεται. 116D υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε όχι. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ψηφοφορία επί της 24. Πέρες τις ψηφοφορίες, εγκρίνεται 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ψηφοφορία επί της 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβαστικής 1. Πέρας. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές, έλεγχος, άρχεται η ψηφορία επί της ε, τροπολογίας 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταλαβαίνω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά σας παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Ε, διαφορετικά θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για κάθε τροπολογία. Τροπολογία 3. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχιτη ψηφοφορία επί της 31. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία επί της 35, πέρες, απορρίπτεται. 36, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά έλεγχος ε, ε, άρχεται η ψηφορία επί της 37 πέρας εγκρίνεται 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία επί της 41. Πέρας και απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία επί της 42. Πέρας. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία επί της 44. Πέρας. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 45. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 Μάλλον την ίδια τύχη με τη 45 θα έχει. Α, ή μάλλον καταπίπτει εξαιτία τη 44. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία της συμβαστικής 3. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος επί της συμβαστικής 6. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 66, 67 και 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για τις τρεις τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 68, δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτή καταπίπτει. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε. Ψηφίζουμε επί της ε, συμβαστικής 7. Ναι, εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84, ε, αυτή καταπίπτει και η 85 καταπίπτει, είναι όμοιες και η 86 καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν στην ε, τροπολογία 127D υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Ψηφίζουμε επί της 127D, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για αυτή την επικοδομητική ψηφοφορία. Σας παρακαλώ, ε, μην κάνετε φασαρία άμα ε, φεύγετε. Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί φεύγετε, σας παρακαλώ όμως, κάντε ησυχία. Λοιπόν, μια και αποφασίσαμε για την αλλαγή της ημερήσιας διάταξης, ε, το σημείο 11 θα εξεταστεί τελευταίο. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως με το σημείο 12, το σημείο 13 και... Αυτά, τα δύο πρώτα. Okay. Ξεκινάμε λοιπόν με το θέμα για την Σιγκαπούρη. Ο David Μάρτιν νομίζω είναι εισηγητής. Thank you, Baron. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μία επικαιροποίηση λοιπόν σχετικά με την εξέταση των τροπολογιών. Σας παρακαλώ ησυχία, λέει ο Πρόεδρος. I'm almost scared to speak myself now. <laughs> Τώρα φοβάμαι να μιλήσω, κι εγώ ο ίδιος. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες. 116 ε, συνολικά λάβαμε. Φυσικά δεν θα τις εξετάσω όλες μία προς μία. Θα επικεντρωθώ σε τέσσερις τομείς που φάνηκαν από τις τροπολογίες. Πρώτα, θέματα φορολόγησης. Ορισμένες τροπολογίες αναφέρονται στο ότι η Σιγκαπούρη είναι φορολογικός παράδεισος. Αυτό δεν είναι σωστό. Ορισμένες ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλιστα έχουν πολύ πιο χαλαρή φορολογική νομοθεσία από τη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα με ε, φυσιολογικό ε, φορολογικό καθεστώς. Έχει λάβει καλή βαθμολογία από το Φόρουμ για την διαφάνεια και την φορολογία για το 2018, όπως και η Σουηδία, η Φιλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία. Έπειτα, ούτε βρίσκεται σε μαύρη λίστα, ούτε βρίσκεται υπό παρακολούθηση σχετικά με τις εφορολογικές της πρακτικές. Η Σιγκαπούρη το 2017 υπέγραψε ε, την Πολυμερή Συμφωνία για τις Αρμόδιες Αρχές σχετικά με την εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς και κοινοποίησε τις προθέσεις της στον ΩΣΑ για την αυτόματη ενεργοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή με όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία δεν είχε συνάψει διμερείς συμφωνίες. Η δέσμευση της Σιγκαπούρης ήδη αναφέρεται στην συμφωνία ε, συνεργασίας. Δεν συμφωνώ λοιπόν με τις τροπολογίες που θέλουν να, που κατανομάζουν την Σιγκαπούρη ως έναν φορολογικό παράδεισο. Το λιμάνι της ε, Σιγκαπούρης είναι πολύ σημαντικό. Η Σιγκαπούρη είναι ένα τεράστιο οικονομικό κέντρο. Σε περίπτωση οικονομικής κρίσης που συζητήθηκε την ε, προηγούμενη φορά, έχουμε τη δυνατότητα να υιοθετήσουμε κατάλληλα μέτρα που θα προστατεύσουν είτε τους επενδυτές είτε τους καταθέτες και θα διασφαλίζουν την ακαιρεότητα και τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Ε, δεν βλέπω λοιπόν κάποιον κίνδυνο πρόκλησης ε, οικονομικής κρίσης ε, όπως αναφέρονται οι τροπολογίες. Και αν δώσουμε το λόγο και στον πρόεδρο τη Επιτροπή, νομίζω και αυτό θα μπορέσει να μα εξασφαλίσει γι' αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι γεωγραφικέ ενδείξει προσφέρονται αυτό, προσφέρεται αυτόματη προστασία σε όλες τις ε, προστατευμένες γεωγραφικές ενδείξεις. Η διαδικασία καταχώρησης όμως θα διεξαχθεί από τη στιγμή που δώσετε στην κατάθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πεπισμένος ότι περισσότερες γεωγραφικές ενδείξεις, αν όχι όλες, θα ε, προστατεύονται και θα ήθελα να, εξασφαλί... να διαβεβαιώσω τους ε, συναδέλφους για το ότι η διαδικασία καταχώρησης στην Σιγκαπούρη είναι ε, δρομολογημένη. Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση για την βιώσιμη εμπορική ανάπτυξη και τη σύμβαση με, το διεθνή, τη Διεθνής Οργάνωση Εργασία. Ε, η Σιγκαπούρη έχει καταγγείλει τις, ε, την, την εξαναγκαστική εργασία και έχει υπογράψει σχετικές συμβάσεις Συμφωνώ και θα στηρίξω τις τροπολογίες όμως που αναφέρουν ότι περιμένουμε μία ένδειξη από τη Σιγκαπούρη για να ε, εισέλθει σε βαθύτερο διάλογο για τα κεφάλαια αυτά και σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη συμφωνώ ότι δεν ε, γίνεται να εφαρμοστεί 100%. Αναμένουμε μία αναθεώρηση το συντομότερο μέσω της ε, ρήτρα αναθεώρησης έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό κυρώσεων ε, ως ε, τελευταία λύση. Ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση για όλα αυτά τα σημεία, τα οποία και εσείς συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε πως είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα μου. Οι δεσμεύσει είναι αξιόπιστες μόνο όταν υπάρχει και ένας αξιόπιστος μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Να ευχαριστήσω ξανά όλους τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους ε, και προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές και στις συμβαστικές τροπολογίες που θα ε, δημιουργήσουμε. Μέχρι τώρα η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Σας ευχαριστώ πολύ. Το, το λόγο θα πάρουν οι σκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Κέλλη Λίπη, ο κύριος Καμάλ επίσης. Η Νάντια Χίρς θα αντικαταστήσει τον κύριο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λίγα λόγια θα πω εξ ονόματος του κυρίου Ατρεμόσα, ο οποίος δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί γιατί βρίσκεται στην Ουάσιγκτον με την ε, επίσημα αντιπροσωπεία ε, του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ήθελα να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στο θέμα αυτό. Λίγες είναι οι τροπολογίες που έχει καταθέσει διότι θεωρεί πως το σχέδιο έκθεση είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτον, θα ήθελε να προσθεθεί ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένη με την ε, συνεργασία που έχει δείξει η Σιγκαπούρη παρά τις καθυστερήσεις από τη δική μας πλευρά. Μετά να αφαιρεθεί αναφορά σε μηχανισμό κυρώσεων. Αυτό δεν μπορεί να το στηρίξει η ομάδα των ε, φιλελευθέρων. Αλλά είναι πεπισμένος ο κ. Σοτρεμόσα ότι η λύση που θα βρεθεί θα είναι κατάλληλη. Το σημαντικό είναι να δώσουμε το πράσινο φως στη συμφωνία αυτή έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο και σε ό,τι φορά την ε, επενδυτική συμφωνία ελπίζουμε να βρεθεί γρήγορα μια λύση η οποία και θα τονίζει τη σημασία της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης αλλά θα ε, διατηρεί τον εθελοντικό της χαρακτήρα, κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια πολύ καλή βάση έτσι ώστε να καταλήξουμε σε δύο δυνατά ψηφίσματα που θα δείξουν την ε, συμφωνία μας και προσβλέπουμε επίσης την καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τους υπόλοιπου κοιόδης. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Άννα Μινέρ, εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω τις ανησυχίες που έχω για αυτήν την συμφωνία η χρηματοοικονομική αγορά της Σιγκαπούρης είναι υπέρ των δέων φιλελεύθερη. Η Σιγκαπούρη έχει πάρα πολλές εταιρείες βιτρίνες και λειτουργεί ως ε, φορολογικός παράδεισος. Αυτό δεν είναι μια φρημένη έννοια, αυτό είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος που ε, κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε μια οικονομική κρίση. Οι χαμηλότεροι δασμοί δεν... Ε, πρέπει να σημαίνει και ότι βέβαια η χώρα είναι φορολογικός παράδεισος, όμως είναι πολύ σημαντικό να δοθούν εγγύησει στα κράτη-μέλη για το ότι θα υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορία και σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο για τους δασμούς. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι πρωτού έχει κυρωθεί η συμφωνία, αλλά δεν συμφωνούμε με το ότι παραβλέπονται τα σοβαρά ζητήματα του περιβάλλοντος ε, της, ε, των ζώων και των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σούλου, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα πάρω τον λόγο εξ ονόματος της κυρίας ε, Μπεγκίν που βρίσκεται σε αποστολή στην ε, Ουάσιγκτον. Όπως και άλλες συμφωνίες και τούτη εδώ με τη Σιγκαπούρη ε, προβλέπει προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Έχει δε αποδεχθεί η Σιγκαπούρη ε, ένα σχετικό ε, μητρό. Όμως προβληματιζόμαστε γιατί αυτό το μητρό δεν έχει ακόμα θεσπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν το γεγονός αυτό, ίσως κάποιες, γεωργικές, συγγνώμη, κάποιες γεωγραφικές ενδείξεις δεν θα αναφερθούν σωστά. Επίσης θα υπάρξει επίσης και ένα τέτοιο σκέλος διοικητικό το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα. Και ένα ακόμα πιο σοβαρό θέμα είναι το εξή. Πριν από λίγο καιρό μάθαμε ότι περίπου 15 γεωγραφικές ενδείξεις ενδεχομένως δεν θα προστατευτούν καθόλου. Μεταξύ αυτών υπάρχουν κάποιες που αφορούν τη χώρα μου, ακόμα ε, περιλαμβάνεται και η Φοντίνα. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, σοβαρό. Επίσης, ε, το γεγονός ε, της έλλειψης διαφάνειας απέναντι στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία μόνο τελευταία πληροφορήθηκε κάποια στοιχεία και ότι η αρχή έγινε το 2013 μέσω απλής επιστολής και μάλιστα την εποχή που ήταν προηγούμενη θητεία και άλλοι ήταν οι υπεύθυνοι βουλευτές. Εμείς θα θέλαμε να ζητήσουμε να μας μεταφερθεί ο πλήρης κατάλογος των γεωγραφικών ενδείξεων που θα προστατεύονται από τη Συμφωνία. Ευχαριστώ. Στην κυρία Μάρτιν Πράτ θα δώσω το λόγο τώρα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την εξαιρετική του, ε, ε, τις εξαιρετικές του γνωμοδοτήσεις όσον αφορά τα δύο θέματα που μας απασχολούν και για την προσωπική του δέσμευση όσον αφορά την αντιμετώπιση των θέματων αυτών. Ο εισηγητής ζήτησε περισσότερες ε, κάποιες ε, πληροφορίες και ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χρηματοδοτικές υπηρεσίες και επίσης το θέμα το οποίο μόλις αναφέρθηκε, δηλαδή το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς τι κάνουμε ακριβώς σε μια FTA όσον αφορά την απελευθέρωση των υπηρεσιών και τι δεν κάνουμε, τι δεν προβλέπεται σε μια ε, συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών δεν τροποποιούμε την ισχύουσα κατάσταση για ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ παλιά ιστορία. Δεν υπάρχει επιπλέον απελευθέρωση ε, ούτε όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων ε, ούτε και όσον αφορά κεφάλαια που προκύπτουν από, τα τις χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές. Ε, απλώς καλύπτουμε τις ε, ε, υποχρεώσεις τις οποίες ήδη έχουμε όσον αφορά τη συνθήκη λειτουργίας αλλά και όσον αφορά και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συμφωνίες με τον ΩΣΑ. Αντιθέτως, σε αυτήν την εμπορική συμφωνία επαναλαμβάνουμε ε, το θεμητό της θέσπισης ε, δημοσίων ε, στόχων. Και είναι γεγονός ότι εμείς δεν προβάλλουμε καμία άλλη απέτηση όσον αφορά ιδιαιτέρως το χρηματοπιστωτικό τομέα. Θέλουμε να συνεχίσει η επιτήρηση, αλλά με τρόπο μη διακριτικό να μην προκύψουν δηλαδή διακρίσεις. Ε, επίσης δεν υπάρχει ε, νομοθεσία χρηματοπιστωτική, δημοσιονομική που θα πρέπει είτε να περιοριστεί είτε να τροποποιηθεί από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επομένως νομίζω ότι είναι σαφές όταν λέμε ότι οι διατάξεις ε, του, της συμφωνίας μπορούν να θεωρηθούν ουδέτερες όσον αφορά προβλήματα ή χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επίσης, ε, μέσω της ε, συμφωνίας μπορεί να επιτευχθεί στενότερη ε, συνεργασία ανάμεσα στους ρυθμιστές από ευρωπαϊκής πλευράς και την ε, Σιγκαπούρη. Όσον αφορά τώρα τον προληπτικό έλεγχο, ε, πάντα ε, ενσωματώνουμε και ένα κεφάλαιο για προληπτικό έλεγχο, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα οι ρυθμιστές, οι ρυθμιστικές αρχές να πάρουν μια σειρά από μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις και στην PCO τη Σιγκαπούρη. Επίσης, ε, πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να δείξω το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Ε, είναι θεμελιώδους ε, σημασίας και οπωσδήποτε δεν είναι σωστό να λέει κανείς ότι δεν αντιμετωπίστηκαν με σοβαρότητα. Οπωσδήποτε η θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας είχε ως ε, προϋπόθεση τον σεβασμό από την πλευρά της Σιγκαπούρης των γεωγραφικών ενδείξεων. Και ευελπιστούμε ότι μετά την έγκριση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σαφές ε, ότι οι ε, αρχές της Σιγκαπούρης θα αρχίσουν τον, τη δέσπιση του καταλόγου βάσει του οποίου θα προκύψει η προστασία των ε, γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν προσαρτηθεί ε, στην συμφωνία. Είναι γεγονός ότι οι χώρες ε, αυτές, όλες οι χώρες στη διάρκεια των συμφωνιών και των διαβουλεύσεων σε επίπεδο Συμβουλίου πάντοτε προστάτεψαν τις γεωγραφικές ε, ενδείξεις ε, και πρέπει να σας πω ότι εμείς διασφαλίζουμε και προσέχουμε έτσι ώστε όλη αυτή η διαδικασία να προχωρήσει με τρόπο ικανοποιητικό και ώστε η τελική συμφωνία και το αποτέλεσμα να είναι ε, ικανοποιητικά για όλες τις χώρες. Πρέπει να σας πω ότι η συμφωνία με την Σιγκαπούρη θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά την σε παγκόσμια παγκόσμιο επίπεδο προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Ε, επομένως, φρονώ ότι ε, η συμφωνία όταν και εφόσον επιτευχθεί θα είναι πολύ ικανοποιητική. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Ο κύριος Καμάλ. Όχι, μετά από σας, αλίμονο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όχι, εντάξει, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Να επαναλάβω βέβαια σε αυτά που άκουσα από την εκπρόσωπο τη ΓΚΟΕ ότι συνήθω αυτή την επιτροπή χρησιμοποιούμε του διεθνεί ορισμού των πραγμάτων. Και μια που αναφέρθηκε προηγουμένω, ε, κοίταξα όλου του διεθνεί οργανισμού και τι λένε για την φοροαποφυγή και του φορολογικού παραδείσου. Σε Σιγκαπούρη δεν είναι σε καμία μαύρη λίστα, σε καμία λίστα ε, ελέγχου, δεν χαρακτηρίζεται ω φορολογικό παράδεισο. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πω ήταν λάθο αν την χαρακτηρίζαμε ω τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν παραμένω πιστό στην άποψή μου, δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την τροπολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ασχολήθηκε με το θέμα τη ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύμβαση τη Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία, θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε τη Σιγκαπούρη να την ε, υπογράψει. Και κατανοώ τι είναι κυρία Μπεγκίνε για τις γεωγραφικές ενδείξεις και εγώ απογοητεύτηκα κάπως από την διαδικασία παρά ε, το ότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, καταβάλει προσπάθειες. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Σιγκαπούρη δεν αναγνωρίζει καμία γεωγραφική ένδειξη και πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Σε αντίθεση λοιπόν με τις άλλες συμφωνίες που απλά είχαμε ένα κατάλογο του, τον δίναμε και τον δέχονταν, η Σιγκαπούρη πρέπει να δημιουργήσει μηχανισμό αναγνώρισης γεωγραφικών ενδείξεων. Είμαι αισιόδοξο ότι όταν δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός θα αναγνωριστούν όλες σχεδόν όλες οι γεωγραφικές ενδείξεις. Όμως ε, υπάρχει, δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο μηχανισμός, υπάρχουν τέλη που πρέπει να καταβληθούν κτλ. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή. Νομίζω πάντως ότι στο τέλος όλης της διαδικασίας θα απολαμβάνουν προστασίες οι γεωγραφικές ενδείξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για τα σημεία 12 και 13. Το ψήφισμα θα εγκριθεί τον Ιανουάριο, οπότε θα δώσουμε και την ε, συγκατάθεσή μας για να προχωρήσουν. Το σημείο 13 ε, έχει να κάνει με την άλλη πλευρά, με τις επενδύσεις. Ντέιβιντ, έχεις πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε 95 τροπολογίες και είναι δυσκολότερο να τις σχολιάσω ή να προσπαθήσω να βρω συμβαστικέ λύσει, ακριβώ διότι αυτέ οι τροπολογίε είτε εκφράζουν την πλήρη στήριξή του ε, στις πολυμερείς Ε, στο δικαστήριο, στο επενδυτικό δικαστήριο, ή ε, θέλουν ένα σύστημα μόνο για τους επενδυτές. Να σας πω επίσης ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών επενδυτή και κράτους δεν υπάρχει πια, τον έχουμε αντικαταστήσει με κάτι πολύ καλύτερο. Και ε, πράγματι η Σιγκαπούρη ποτέ δεν είχε αναγκαστεί να προσφύγει σε μηχανισμό επίλυση διαφανών επενδυτή και κράτους. Όμως, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, υπάρχουν 13 κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει διμερείς ε, συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη και το επενδυτικό. Και το επενδυτικό αυτό δικαστήριο θα αντικαταστήσει αυτές ε, τις ε, συμφωνίες. Αυτό που θεωρούμε λυπηρό είναι ότι δεν υπάρχουν διατάξεις για τις υποχρεώσεις των επενδυτών και δεν υπάρχει μηχανισμός προσφυγής για την περιπτώση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι σημαντικό για τη δική μου πολιτική ομάδα, όμως ε, θα αφήσω την Επιτροπή να το συζητήσει πριν προτείνουμε διάφορα, διάφορες δικές μας ε, ιδέες για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας. Έχω γενικά εκπλαγεί από τις ε, που είδα τον Οκτώβριο. Το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει με μεγάλη πλειοψηφία την στήριξη των ε, πρωτοβουλειών ε, προστασίας. Και θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω τους εσκαιώδεις εισηγητές και ελπίζω πως γρήγορα θα βρούμε συμβαστικέ λύσεις, αν και γι' αυτό το θέμα θα είναι πιο δύσκολο. Ο κύριος Καμάλ έχει το λόγο για τους σκιώδεις ηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε έναν κύκλο συζητήσεων για το θέμα αυτό. Ορισμένοι αναρωτήθηκαν μάλιστα γιατί χρειάζεται προστασία των επενδυτών έτσι και αλλιώ, γιατί οι μεγάλε εταιρείε να έχουν μεθόδου προσφυγή και δίχτυ προστασία. Αυτό το έχουμε συζητήσει και στη δική μα ε, ομάδα. Υπήρξαν ε, συνάδελφοι που δεν θεωρούσαν καθόλου κατάλληλο το μηχανισμό επίλυση διαφορών επενδυτή και κράτου, πω θέλαν περισσότερη διαφάνεια. ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Νομίζω όμως ότι για την δική μας ομάδα το βασικό είναι να τελειώνουμε. Και εμείς βιαζόμαστε όπως όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρω πως ο Ντέιβιντ έχει κάνει κάποιες ε, σχετικές συζητήσεις, προσπαθεί να ε, ξεπεράσει τα εμπόδια αλλά να πω ότι για όσους έχουν ασκήσει κριτική στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή και κράτους, το νέο σύστημα είναι πολύ ε, καλύτερο. Χαρακτηρίζεται από περισσότερη ε, διαφάνεια. Αυτό όμως που πρέπει να, ε, να δούμε είναι αν, αν χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα γενικότερα και εάν πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ για να δημιουργηθεί ε, νομικό προηγούμενο. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μινέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύρια Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση έρχεται πολύ νωρίς, μιας και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης μπορεί να λάβει αποφάσεις και να γνωμοδοτήσει σχετικά με αυτή τη συμφωνία και την προστασία των επενδύσεων. Εμείς προτείνουμε λοιπόν να ε, λάβει χώρα αργότερο έλεγχος αυτού του κειμένου. Ε, το σύστημα των επενδυτικών δικαστηρίων είναι το ίδιο με αυτό που υπάρχει. Υπάρχει αυτό το ρυθμιστικό πάγωμα που περιορίζει τα δικαιώματα των νομοθετών, των κυβερνήσεων, ε, αντίθετα με αυτά των επιχειρήσεων. Όποιο και αν είναι το σύστημα δεν επιτρέπει σε ΜΚΟ και συνδικάτα να παρέμβουν στη διαδικασία. Εμείς πιστεύουμε ότι τα τοπικά δικαστήρια πρέπει να ε, αποφανθούν και στη συνέχεια θα υποβάλουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι από τους βουλευτές που υπέβαλαν τροπολογίες ε, κατά αυτής της πρότασης, για πολύ απλούς λόγους. Δυστυχώς, στη πολιτική δεν ακούμε συχνά για ε, βασική, ουσιαστική δικαιοσύνη. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να δοθούν ε, δικαιώματα σε όσους έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση και απ' την άλλη να επιβαρύνονται οι κοινότητες, οι εργάτες, όσοι επηρεάζονται αρνητικά περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να δημιουργηθεί ένα παράλληλο δικαστικό σύστημα για τις επιχειρήσεις και το γεγονός ότι υπάρχουν παρεμβάσεις στο σύστημα και όπως είπε η κυρία Μινέρ, ε, ε, γίνονται προσπάθειες ε, βελτίωσης, ε, δημιουργεί αδυναμίες και άνηση μεταχείριση απέναντι στον νόμο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαι κατά της Συμφωνίας Προστασίας των Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μία ε, συμφωνία προστασίας ε, ε, επενδύσεων χωρίς αρνητικό αντίκτυπο. Δεν μπορεί να αντικατασταθούν οι διμερείς συμφωνίες χωρίς τη σύσταση δικών δικαστηρίων. Δεν ήταν όμως τέτοια η πρόθεση στις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, ο λόγος είναι χρηματοοικονομικός. Δεν υπάρχει σύνδεσμος ανάμεσα στις επενδυτικές ροές και την επίλυση των διαφορών. Είναι ξεκάθαρο και από μελέτες ότι μπορούν να προαχθούν οι επενδύσεις χωρίς τη σύσταση ειδικών δικαστηρίσεων δεν υπάρχει σχέση. Δεν υπάρχουν οικονομικοί λόγοι για να συσταθούν τέτοια ειδικά δικαστήρια. Τρίτος λόγος, υπάρχει θέμα ε, χρηστής διακυβέρνησης. Περιμένουμε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, αποφανθεί για το αν μια τέτοια συμφωνία είναι συμβατή με την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Άρα αυτό που υπόθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση όταν ε, ψηφίσαμε για τη συμφωνία ΣΥΤΑ και ε, ε, περιμέναμε, δεν, καθυστέρησε η ψηφοφορία και περιμέναμε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές ε, πιθανότητες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει αρνητική απόφαση κατά της ε, συμφωνίας αυτά, αυτής. Υπάρχουν λοιπόν δύο διαφορετικές συμφωνίες και πρέπει να γίνουν διαφορετικές ε, ψηφοφορίες. Εγώ λοιπόν θα ψηφίσω κατά αυτής της ε, συμφωνίας, γιατί στόχος δεν είναι να δημιουργηθούν αρνητικοί κανόνες σχετικά με τη διακυβέρνηση. Ε, θέλετε να λάβετε το λόγο και ε, σχετικά με τη Σιγκαπούρη. Χαίρομαι για τη δουλειά που επιτέλεσε ο κύριος Μάρτιν. Τον ευχαριστώ γι' αυτό. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Έχουμε, έχουμε υποβάλει τροπολογίες. Η Σιγκαπούρη πρέπει να τηρεί τις ίδιες θεμελώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο ένας προορισμός των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι η συμφωνία αντικαθιστά διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και Χαιρετίζω αυτή την ε, ε, συμφωνία. Η συμφωνία αυτή περιέχει τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των επενδύσεων και υπάρχουν διατάξεις που δεν προβλέπονται στις διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τη Σιγκαπούρη. Σε ό,τι αφορά το σύστημα ε, ειδικών δικαστηρίων. Αναφέρθηκε το προηγούμενο με τη Συμφορία Ελεύθερων Συναλλαγών με το Καναδά. Είναι σημαντικό να προστατευτούν οι επενδυτές με διαφανή τρόπο και να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων μας. Είναι... Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι προϋποθέσεις ε, σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούν οι επενδυτές να προσφύγουν στο δικαστήριο Θα είναι ε, σημαντικό αυτά τα δικαστήρια να διασφαλίσουν την ασφάλεια δικαίου. Να συνεχίσω. Μακροπρόθεσμος στόχος, η θέσπιση ενός διεθνούς ε, συστήματος δικαστηρίων. Γι' αυτό και καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία σύστασης ε, ειδικών δικαστηρίων για την επίλυση εμπορικών διαφορών. και νομίζω ότι το υποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό. Σε ό,τι αφορά το TTIP, ε, νομίζω ότι έχουν γίνει θετικά βήματα. Ε, είναι σημαντικό να διασφαλιστούν ε, τα, η βιώσιμη ανάπτυξη, τα δικαιώματα των ε, εργατών, θέματα ε, χρηστής διακυβέρνησης κτλ. Όπως έχουμε πει, πιστεύω ότι αν δεν ε, συμφωνήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα, τα συμφέροντα των επιχειρήσεών μας σε ό,τι αφορά το ελεύθερο εμπόριο. Είναι σημαντικό να καλύψουμε το χάσμα. Δεν υπάρχει λόγος να απορρίψουμε αυτή την πρόταση. Είναι θετικό να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά υπόθησαν και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μια ερώτηση που επανέρχεται διαρκώς. Ε, γιατί ε, πρέπει να έχουμε προστασία, συγγνώμη, συμφωνία προστασίας ε, επενδύσεων με την Σιγκαπούρη. Πρώτον, να σας πω ότι δεν ξεκινούμε από κενό και από λευκή σελίδα. Έχουμε μια, ένα ολόκληρο σύστημα ε, επενδυτικής πολιτικής ε, και συμφωνιών για επενδύσεις που έχει ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια. Ε, και το Συμβούλιο και η Κομισιόν προσπαθεί να βελτιώσει, να τροποποιήσει αυτό το πλαίσιο. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι θέλουμε να αντικαταστήσουμε ε, τις 13 μεμονωμένες διμερείς που έχουν, συμφωνίες που έχουν με τη Σιγκαπούρη Ορισμένε χώρε με μία που θα ισχύει για όλους. Δεύτερον, η Σιγκαπούρη μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλε συμφωνίε που είτε ε, διαπραγματευόμαστε είτε πρόκειται στο μέλλον να διαπραγματευτούμε στην ε, περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, χώρες ΑΣΕΑΝ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να μην ε, υποτιμάτε παρακαλώ την μεγάλη σημασία που μπορεί να έχει για μελλοντικές συμφωνίες αυτή η συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Επίσης, ε, μέσω της συμφωνίας αυτής ε, θα προκύψει να ε, ε, ε, μια ισορροπία γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινούμε όλοι από το ίδιο σημείο είτε μιλάμε για την Κίνα είτε μιλάμε για την Ιαπωνία είτε τον Καναδά όσον αφορά τις συμφωνίες και βεβαίως οπωσδήποτε βασιζόμαστε και για τις συμφωνίες αυτές είτε στη συνολική προοδευτική εταιρική σχέση του ειρηνικού CPTPP είτε άλλες ε, συμφωνίες ε, επίσης ε, θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι. τούτο εδώ είναι ένα απαραίτητο βήμα. Είναι μία εκ των ουκάνευ προϋπόθεση έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς να δημιουργήσουμε πολυμερή επενδυτικό, πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο στο μέλλον ε, η επίλυση διαφορών ε, ε, επενδύσεων μπορεί να είναι πολύ μεγάλες και δεν μπορούμε να έχουμε ένα ικανοποιητικό βαθμό αντιμετώπισης αυτών των διαφορών εάν δεν μπορέσουμε να κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα. Και να πούμε επίσης ότι και η Σιγκαπούρη αναλαμβάνει δεσμεύσεις ε, απέναντί μας, έτσι ώστε δεσμεύεται δηλαδή για αυτό το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο. Όταν ε, θα ψηφιστεί το IPI εδώ και στην Ολομέλεια, παρακαλώ πολύ σκεφτείτε τα όλα αυτά και ίσως ε, αποφασίσετε ότι αξίζει να προωθήσετε ένα σύστημα προστασίας ε, το οποίο έχει δώσει την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν πολλά ευαίσθητα θέματα και όσον αφορά την διαφάνεια και όσον αφορά την έλλειψη προσφυγών ε, και όσον αφορά τους δείκτες ε, και που αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα προς ένα πραγματικά πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 1.400 διμερείς ε, επενδυτικές ε, συμφωνίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό θα είναι αυτό το πρώτο βήμα. Ακόμα και αν ε, όμως ε, καταψηφίσετε την ε, συμφωνία, δεν θα εξαφανιστούν οι επενδυτικές συμφωνίες. Θα επαναδιαπραγματευτούν, θα αλλάξουν λίγο, θα ξανασυμφωνηθούν. Δεν πρέπει να εξαφανιστούν. Ελπίζουμε βέβαια ότι εσείς θα επιλέξετε την πρώτη επιλογή, δηλαδή θα δώσετε το πράσινο φως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και βεβαίως εμείς όλοι ελπίζουμε ε, ότι η νέα προσέγγιση βασίζεται στην ε, παλιά ε, προσέγγιση. Υπάρχουν ακόμα 200 συμφωνίες οι οποίες διμερείς, οι οποίες ισχύουν ακόμα μεταξύ κρατών μελών. Και νομίζω ότι αυτό το παλιό σύστημα ISDS ε, θέλουμε όλοι ISDS, θέλουμε να το αφήσουμε πίσω μας. Μα την... Ε, σύντομα. Η Ανμαρή Μενιέ ε, δεν είναι ε, ε, και οι σεβονίμων ε, μου καθήμενοι δεν συμφωνούν με τις επενδύσεις. Δεν μπορώ λοιπόν να σας αλλάξω γνώμη, αλλά εάν κάποιος θέλει αυτού του είδους τις επενδύσεις και θέλει οπωσδήποτε προστασία των επενδύσεων, τούτο εδώ είναι το καλύτερο εργαλείο. Μιλάμε για ένα ε, ε, σύστημα επενδυτικ, πολυμερούς επενδυτικού ε, δικαστηρίου το οποίο θα συνάδει με τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα είναι πολύ πιο διαφανές, θα είναι πολύ πιο προστατευτικό Απ' την άλλη πλευρά, εάν δεν συμφωνείτε εξ αρχής με κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να σας προσπαθήσω. Ε, να σας ε, πείσω, συγγνώμη, δεν μπορώ να σας πείσω, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάνουμε, περνάμε στο ε, προηγούμενο θέμα το οποίο το είχαμε αλλάξει. Ε, ενίσχυση ανταγωνιστικότητα εσωτερική αγορά μέσω ανάπτυξη Ελληνική Ένωση κτλ. Είναι το σημείο 11, το τελωνιακό ζήτημα, λέει ο πρόεδρο. Έπρεπε να είναι εδώ ο κύριο Νικόλα Ντάντι, αλλά δεν είναι εδώ, άρα να τα πει ο κύριο Μάρτιν. Λοιπόν, διαβάζω το κείμενό του. Ε, η γνωμοδότηση την οποία συζητούμε αφορά τη διακυβέρνηση της Τελωνιακής Ένωσης. Στο κείμενό μου εστιάζω τις παρατηρήσεις μου σε κάποια πιο σημαντικά ε, ζήματα τα οποία εδώ ε, θα αναφέρω εν συντομία. Πρώτα, πρώτα απ' όλα θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πλήρης εφαρμογή των όσων έχουν υπογραφεί από τον προταθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και έχουν επικυρωθεί από 130 χώρες. Επίσης, πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου αλλά και με τον ΩΣΑ όσον αφορά τα θέματα αυτά. Δεύτερον, Χρειαζόμαστε διασφαλίσεις ε, καλής λειτουργίας ε, των τελωνίων που θα δώσει τη δυνατότητα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα καλύτερο και ενιαίο πρόσωπο όταν διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των αρχών Τελωνιακής Ένωσης, κυρίως στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών. Επόμενο, η προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και των πολιτών είναι ε, σημαντική προϋπόθεση και απορρέει και αυτή από, την, από τον καλό έλεγχο των όποιων προϊόντων κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από ποια χώρα προέρχονται τα αγαθά ή ε, ποιο σημείο εισόδου επιλέγεται. Δεν μπορεί δηλαδή να ε, υποκύψουμε στο forum shopping. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να εναρμονιστούν όσο γίνεται περισσότερο ε, οι τελωνιακές διαδικασίες και να υπάρξουν κοινές, ε, ε, κοινές ποινές για περίπτωση παράβασης. Επόμενο σημείο ε, η είναι ένα, ε, ε, η ψηφιοποίηση είναι σημαντικό στοιχείο και μπορεί να οδηγήσει σε πιο λειτουργικά τελωνία. Επίσης, η ψήφο, ψηφιοποίηση ε, μπορεί να δώσει την ε, δυνατότητα διευκόλυνσης των εμπορικών ε, ροών, κυρίως όσον αφορά προερχόμενους από τρίτες χώρες και βεβαίως την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Επίσης, ε, να υπενθυμίσουμε ότι μετά από, την, ε, από τον Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα. Ε, τρίτη χώρα λοιπόν μετά από την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που θα μεταβάλει και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως επισημαίνουμε ότι η διαδικασία του Brexit δεν πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη ή στην διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι στη διάθεσή σας για ε, τα σχόλιά σας και βεβαίως προσδοκώ σε πλήρη συνεργασία. Σε Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Chair, um, for giving me the floor. Σας ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για την πρόσκληση που μου έκανε να έρθω σήμερα. Όπως ε, γνωρίζετε, έχουμε ήδη συζητήσει στην ε, Επιτροπή Ίνκο, στην παρουσίαση τη σχέδιο έκθεση της κυρίας Ροζιέρ. Έδειξε την πλήρη δέσμευση των κρατών μελών προς μία πλήρη αυτοματοποίηση της Τελωνιακής Ένωσης και αναγνωρίζει την ε, σημασία μίας ε, εύρυθμη τελωνειακής ενωση για την ενιαία αγορά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία περαιτέρω δρομολόγηση ε, του Τελωνιακού Κώδικα περίπου το 90% της τελωνιακής διαδικασίας είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, όμως ο τελωνιακός κώδικας πηγαίνει ακόμα παραπέρα και στόχος του είναι η ενιαία εφαρμογή, η αντικατάσταση των εθνικών προδιαγραφών με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, κάτι το οποίο θα διασφαλίσει και ενιαία αντιμετώπιση ε, των ε, εισαγωγών από τρίτες χώρες τη στιγμή που μπαίνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος και θα αποτρέψει την ε, αναζήτηση ευνοϊκής δικαιοδοσίας. Σε ό,τι αφορά την έκθεση του κυρίου Ντάντι, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη αναπτύσσει ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα εφαρμόζονται οι κανόνες ε, του, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνίων. Αυτό το πλαίσιο συνδυάζει από τη μία σύγχρονους κανόνες, σε διευκόλυνση του εμπορίου, αλλά και περισσότερο ασφαλείς σε διαδικασίες. Να σας πω επίσης ότι και εγώ ήμουν ε, υπάλληλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνίων και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συμμόρφωση προς τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είμαστε πολύ μπροστά. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ντάντι, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τον ε, οργανισμό, να συνεισφέρουμε στο έργο του, να συνεχίσει η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Πρόσφατα παρουσιάσαμε τις ε, διαδικασίες και θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε και άλλες έτσι ώστε να παροτρύνουμε τους εταίρους μας κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, για να θεσπίσουν και οι ίδιοι νέους σύγχρονους κανόνες. Αναφερθήκατε στους ελέγχους και στις μεθόδους ε, για μείωση του διοικητικού άχθους. Αυτή τη στιγμή ε, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνίων αυτό που κάνουμε για να, για να διαχειριστούμε τον κίνδυνο είναι να δημιουργήσουμε εργαλεία τα οποία εστιάζουν στους κακούς εντό εισαγωγικών και που διευκολύνουν το νόμιμο εμπόριο. Γι' αυτό πρόσφατα δημιουργήσαμε ένα κατάλογο κοινών κριτηρίων για την αντιμετώπιση του κινδύνου, έγιναν απλουστεύσεις και τώρα αυτοί οι κανόνες ισχύουν και για τους ε, νόμιμους οικονομικούς φορείς, ανταμείβοντάς τους ε, για την ε, νομιμότητα των εργασιών τους, αλλά και μειώνουν τη γραφειοκρατία. Συνδυάζουμε λοιπόν την αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνου με τις διάφορες απαιτήσει σχετικά με την παροχή δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο, έτσι ώστε στο εμπόριο να μην χρειάζεται να συμμορφωνόμαστε με διάφορα σύνολα κανόνων για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Ε, αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε ναι, βελτιώσεις και επικαιροποίησει των υφισταμένων συστημάτων. Από το 2017 υπάρχει το κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, το οποίο προβλέπει μια στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και υποχρέωση όταν οι έλεγχοι διεξάγονται από τα κράτη-μέλη επιτόπου, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο, να εφαρμόζεται ο τελωνιακό κώδικας και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Δηλαδή, αν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι έρχεται μια ύποπτη εισαγωγή, να ενημερώσει άλλα έτσι ώστε και εκείνα να πράξουν τα δέοντα. Αυτό είναι στο πλαίσιο λοιπόν και του τελωνιακού κώδικα και του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου γίνονται τακτικές συζητήσει και συναντήσει με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αυτή η καλή συνεργασία. Να πω επίση ότι παρά το γεγονός ότι η ευθύνη για του ελέγχου είναι στα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει και η ίδια διάφορες διερευνητικές αποστολές ε, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμών και αν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν σωστούς ελέγχους, τότε λαμβάνονται μέτρα, ξεκινούν ε, διαδικασίες επί παραβάση, αν αυτή η ελέγχη δεν είναι αποτελεσματική, ας πούμε. Κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά, μπορώ να πω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πληροφορική, τα συστήματα πληροφορικής, η μεταρρύθμιση και επικαιροποίηση τους είναι κέρια σημασίας. Αυτό γνωρίζουμε πως είναι δύσκολο, ιδιαίτερα επειδή ξεκινάμε βασισμένοι πάνω σε ένα ισχύον σύστημα. Ο τελωνιακός κώδικας δεν αφορά μόνο την εφαρμογή ναι, και την υλοποίηση νέων συστημάτων, αλλά και την επικαιροποίηση των εφισταμένων για εισαγωγές, εξαγωγές, για διέλευση. Αυτό είναι ίσως και το δυσκολότερο από όλα διότι μιλάμε και για την συνέχεια των συστημάτων. Είναι πιο δύσκολο να αναβαθμίσεις ένα σύστημα που έχει λειτουργήσει σωστά εδώ και πολλά χρόνια από το να χρησιμοποιείς ένα εντελώς καινούριο σύστημα πληροφορικής. Βέβαια, βλέπουμε ότι κατά την εφαρμογή των συστημάτων χρειάζεται να ανταπεξέλθουν σε νέες προκλήσεις, για παράδειγμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εδώ παρουσιάστηκαν διάφορες νέες πτυχές, τις οποίες έπρεπε να χειριστούμε, έτσι ώστε να μην έχουμε έναν τελο, ενωσιακό τελωνιακό κώδικα που ναι μεν χρησιμοποιείται, αλλά δεν είναι σε θέση να το απεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Πρέπει λοιπόν να εναρμονιστεί η λειτουργία του με το μοντέλο του, της Παγκόσμιας ε, Οργάνωσης Τελωνίων. Αυτό είναι μια πρόκληση. Γιατί πρέπει να δούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα γνωρίζετε ίσως πως έχουμε ζητήσει αναβολή και παράταση της προθεσμίας του 2020 για τα συστήματα πληροφορικής. Εδώ και αρκετό καιρό συνομιλούμε με τα κράτη-μέλη και έχουμε καταλήξει σε ένα σχέδιο που θα πάει μέχρι το 2025. Βέβαια είναι στο χέρι των συνομοθετών να αποφασίσουν γι' αυτό, αλλά θα έλεγα ότι κάτι που περιπλέκει την υπόθεση και τα συστήματα είναι ότι υπάρχουν οι ευρωπαϊκές πτυχές αλλά και η διεθνής διάσταση. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε διασυνδέσεις ανάμεσα στα συστήματα έτσι ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία. Και θα συνεχίσει να υφίσταται το εθνικό επίπεδο μαζί με το ευρωπαϊκό, διότι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε την εθνική διάσταση. Γι' αυτό λοιπόν Λέω πως ε, μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουμε μάλλον καταφέρει να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα συστήματα και να είναι μαζί του, μεταξύ τους συμβατά. Νομίζω και κάποιος ευρωβουλευτής στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, κατά την παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Ροζιέρ, είπε ότι θέλουμε το σύστημα να είναι καλό. Δεν θέλουμε να βιαστούμε και να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι επικαιροποιημένο, δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτά που πρέπει να κάνει. Όταν μπλοκάρει ένα σύστημα, δεν μπορεί να γίνει μια εισαγωγή. Και αναφέρετε κι εσείς ο ίδιος ότι στο πλαίσιο του Brexit ε, θα υπάρξουν προβλήματα. Όμως, να, διασφαλίσω και, να, να διαβεβαιώσω και τον εισηγητή και τους ε, υπόλοιπους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει τους κανόνες του Ενωσιακού Τελωνιακού Κώδικα και την σχετική νομοθεσία αλλά και επίση ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ο David Μάρτιν έχει το λόγο χρειάζεται νομίζω να σχολιάσω. Να ευχαριστήσω πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ε, πολύ καλά και λεπτομερή της σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Τώρα περνάμε στα σημεία 16 και 17 οι συμφωνίε με την σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Ο κύριο Ζεχραντήλ είναι ο εισηγητή, δυστυχώ απουσιάζει. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπάνερμαν, ο οποίο τον αντικαθιστά. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, μιλώ εξ ονόματο του κύριου Ζεχραντήλ. Όπω γνωρίζετε, ο κύριο Ζεχραντήλ προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Πήγα και εγώ σε αυτές τις ε, συναντήσεις που έχουν γίνει στο Βιετνάμ και ο κύριος Ζαχραντήλη θα ήθελε να πει ότι η διαδικασία αυτή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012, ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015 σε πρώτο στάδιο, έτσι ώστε να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για την Σιγκαπούρη και ε, κατόπιν αυτού διαχωρίστηκε η συμφωνία σε εμπόριο και επενδύσεις. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την ε, διαδικασία εντός της ε, παρούσας και να υπογράψει τη συμφωνία. Η Αυστριακή και η επερχόμενη Ρουμανική Προεδρία έχουν δεσμευτεί να προσπαθήσουν το καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν τους ε, επικροτούμε γι' αυτό. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για το ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί η συμφωνία τώρα, εντό τη θητεία. Πρώτον, γιατί θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη στο Βιετνάμ και στι ε, εταιρείε Ευρωπαϊκή Ένωση που δραστηριοποιούνται εκεί. Ε, θα έχει πρόσβαση σε μια δυναμική περιοχή στην Νοτιοανατολική Ασία και σε χαμηλό κόστο παραγωγή. Και επίση θα, θα ανοίξει μια νέα αγορά για εξαγωγέ. Θα βοηθήσει επίση η συμφωνία αυτή ε, την πρωτογενή αγορά του Βιετνάμ κατά 15% του ΑΕΠ του. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ελπίζουμε να είναι διαθέσιμο στην επόμενη ε, συνάντηση. Αυτό τουλάχιστον έχουμε ζητήσει. Τώρα, δεύτερο στοιχείο. Αυτή η συμφωνία είναι ένα νέο, πολύ φιλόδοξο μοντέλο εμπορικών συναλλαγών με τις αναδυόμενες οικονομίες θα καταργήσει σχεδόν όλους τους δασμούς, το 99% αυτών και θα απελευθερώσει το Βιετνάμ το 65% ε, των ε, εξαγωγών του, των εισαγωγών του. Η διαδικασία αυτή προβλέπει μια σταδιακή εξάλληψη μέσα σε περίοδο 10 ετών. Είναι λοιπόν ένα καλό μοντέλο αυτό. Τρίτον, προωθεί τι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι καταλήτης για μεταρρυθμίσεις, είναι αυτή η ήπια ε, δύναμη της Ένωση. Εφόσον κυρωθεί η συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει περισσότερη ε, διαπραγματευτική ικανότητα, έτσι ώστε να πιέσει το Βιετνάμ για να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό και για ε, τις ε, πτυχές των εργασιακών δικαιωμάτων. Υπάρχουν οι σχετικές συμβάσεις της Παγκόσμιας Μιας Οργάνωσης Εργασίας. Προβλέπεται συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών. Και τέλος, ο κύριος Ζαχραντή σκοπεύει να μεταβεί στο Βιετνάμ το 2019, πολύ σύντομα. τώρα, Περνάμε στην Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων που είναι ξεχωριστή. Ο κ. Ζαχραντήλη θεωρεί πως είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος επενδυτής στο Βιετνάμ, όπως έχει γίνει και με άλλες ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών έχουν γίνει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή και κράτους και αυτή η συμφωνία είναι η δεύτερη ξεχωριστή συμφωνία που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια τρίτη χώρα. Φυσικά υπάρχουν και τα κατά αυτού του διαχωρισμού, ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να κυρωθεί όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από όλα τα εθνικά ή, σε ορισμένε περιπτώσει, περιφερειακά κοινοβούλια, των κρατών μελών. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει από 2-3 χρόνια, γιατί τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν ε, τη συμφωνία. Αυτά θα ήθελε λοιπόν να πει συνοπτικά ο κύριος Ζαχραντήλ. Ελπίζει να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό μέχρι το τέλος της ε, κοινοβουλευτικής θητείας που διανύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές ο κύριος Μάρτιν πρώτος, εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, μιλώ εξ ονόματος της συναδέλφου που δυστυχώς απουσιάζει, οπότε θα διαβάσω και εγώ τη δήλωσή της όπως μου την έχει δώσει. Η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ έχει ορισμένες θετικές πτυχές για την πρόσβαση στην αγορά, για τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, γεωγραφικέ ενδείξει και τι δημόσιε συμβάσει και έχει τη δυνατότητα ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ. Η συμφωνία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τρεις άλλους ε, λόγους. Πρώτον, είναι η πιο ολοκληρωμένη διμερή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που έχει διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία αναπτυσσόμενη χώρα. Δείχνει ότι τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης δεν είναι μόνο εστιασμένα στο, στον ανεπτυγμένο κόσμο. Δεύτερον, αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για, την, για τις χώρες αυτές και την ανάπτυξή τους, τις χώρες της περιοχής, αλλά και για τις μελλοντικέ συμφωνίες για την ανάπτυξη της περιοχής αυτής. Τέλος, το Βιετνάμ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα λόγω της γεωγραφικής και γεωπολιτικής του θέσης και ελπίζουμε η διαδικασία αυτή να δώσει όθηση όχι μόνο στην ε, οικονομία και στις συναλλαγές αλλά και στην αναγνώριση των κοινών μας αξιών. Η ίδια η συμφωνία είναι αποτέλεσμα εξαιρετικής προσπάθειας από τη διαπραγματευτική ομάδα, όμως το κεφάλαιο για τον πόρο και τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει ακόμα ελλείψεις. Ζητούμε λοιπόν τη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ να συμμορφωθεί με αυτές ε, με τις διεθνείς συμφωνίες. Περιμένουμε λοιπόν από τις αρχές της χώρας ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με το μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να πιστεύεσαι τον ε, εταίρο σου. Γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν έχουν γίνει αρκετά όσα θα έπρεπε για αυτά τα πολύ λεπτά ζητήματα. Η συνάδελφος θα ήθελε επίσης να προσθέσει τα εξής. Πρώτον, θα χρειαστεί σαφής δέσμευση ως προς το χρονοδιάγραμμα, όπως προτού περάσει στην κύρωση. Πρέπει να, το Βιετνάμ να κυρώσει τη Συμφωνία 87, και 105 της Παγκόσμιας Οργανώσης Εργασίας. Επίσης, χρειάζεται να διευκρινιστεί το πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτής της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών και να υπογραφεί η Παγκόσμια Διακήρυξη των ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επίσης υπάρχουν ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την ε, ελευθερία της ε, έκφρασης. Γι' αυτό λοιπόν η Σκιώδη Συγκήτρια θα ήθελα να συνεργαστεί με όλους τους Σκιώδες για να οδηγηθούμε στην γρήγορη υπογραφή της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος του ΕΝΕΦ e έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι εμπορικές συμφωνίες είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικές για την Ευρώπη, διότι διευρύνουν την οικονομία μας. Και η εμπορική συμφωνία του Βιετνάμ σε αυτή την γραμμή εγγράφεται. Για το σκοπό αυτό θα ήθελα να ζητήσω ιδιαίτερη προσοχή ε, στα ζητήματα τα οποία αφορούν την εξαγωγή του ρυζιού ε, όπου πρόσφατα είδαμε για τη Μαϊνμάρ και την Καμπότζη ε, να επικαιροποιείται η ρήτρα διασφάλισης. Άλλο σημείο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, τα οποία συζητήθηκαν ε, και εδώ. Επίσης ε, θέματα όπως η εργασία των ανηλίκων και η προστασία των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εξίσου σημαντικό και τα περιβαλλοντικά πρότυπα π.χ. σε σχέση και με την χρήση φαρμάκων ε, στην γεωργία, ε, την χρήση πλαστικού, γιατί εμείς έχουμε πρόσφατα εγκρίνει ψήφισμα για την κατάργηση της ε, χρήσης πλαστικών ε, μίας ε, χρήσης εδώ, ενώ το 95% της μόλυνσης από πλαστικά προέρχεται στις θάλασσες του, του, του πλανήτη από μερικά μεγάλα ποτάμια, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στην Ασία, όπως ας πούμε ο Μεκόγκ θα πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί μια πολιτική που δεν θα είναι, ε, που, που οπωσδήποτε θα ευθυγραμμίζεται με τις αρχές που έχουμε εμείς θέσει τους εαυτούς μας σε συμφωνία με μια άλλη χώρα, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ε, σέβεται τις αρχές και τους κανόνες που έχουμε θέσει εμείς στον εαυτό μας και θα πρέπει να ελέγχουμε ότι ας πούμε στις ε, χώρες αυτές δεν θα χρησιμοποιείτε το πλαστικό το οποίο μέσω των ε, ε, ποταμιών θα φτάσει στις θάλασσες του πλανήτη. Ευχαριστώ. Thanks lot for the... Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Ανμαρή Μινέρ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Διαπραγματευόμαστε μία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Βιετνάμ, ενώ υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Πρόκειται για αναπτυσσόμενη χώρα και δεν μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς GSP+, στο ειδικό καθεστώς. Μία ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου εστιάζει λιγότερο σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατάσταση των τρομήνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ είναι πολύ ανησυχητική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, ξέρει ότι πρόκειται για ε, θεμελιώδεις αξίες. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. συστάθηκε η σύσταση ομάδας είναι κάτι πολύ περιορισμένο αφού δεν ε, γίνεται ε, δεν υπάρχει ελεύθερη έκφραση θα γίνει αυτή η χώρα όπως το Μπαγκλαντές που εστιάζει στην εξαγωγή κλαστοϊφαντουργικών ε, ειδών δεν είναι αυτό που θέλουμε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συμφωνία είναι πολύ σημαντική. Συζήτησα με τον εισηγητή για το χρονοδιάγραμμα και υπόθηκε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωμοδοτήσουν άλλες επιτροπές, αλλά το χρονοδιάγραμμα δεν μας επιτρέπει κάτι τέτοιο και θεωρώ ότι είναι κρίμα. Κυρίως δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα ψηφίσει το Συμβούλιο. Είναι πολύ λοιπόν στενά τα περιθώρια και οι προθεσμίες. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ε, Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με το Βιετνάμ. Ως μέλος της ομάδας θα σας καλέσω να εστιάσετε στο κεφάλαιο που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί υπάρχει μία συσχέτιση ανάμεσα στο εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, η συμφωνία αναφέρεται ότι κάθε χώρα πρέπει να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος, των ε, δασών και των καλλιεργειών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την σύναψη εθελοντικών ε, συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου και σε αυτή την, κατάσταση, την περίπτωση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μία ε, εθελοντική συμφωνία ε, εταιρικής σχέσης μπορεί να συμβάλλει στις εξαγωγές μιας χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζοντας την προέλευση των προϊόντων. Και θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την προστασία των επενδύσεων. Η ομάδα μου πιστεύει ότι πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμβατότητα ανάμεσα στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ε, με το Καναδά και ε, τις ε, διεθνείς συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, ενθαρρυντικά αυτά που λένε οι συνάδελφοι. Όπως και για τη Σιγκαπούρη, έχουμε μεγάλες προπτικές ε, με τις χώρες της ε, Ασίας και το Βιετνάμ ανήκει σε αυτές. Επισκέφτηκα αυτή τη, χώρα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πάνω σε διάφορα ε, ζητήματα που έχουν προκύψει. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Δεν αλλάζουν αυτά τα ζητήματα εν μια νυχτή. Μία οικονομία που αναπτύσσεται έχει θετικές συνέπειες για όλους. Ε, φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ουσιαστικό ζήτημα. η μία συμφωνία με το Βιετνάμ θα μπορούσε να ε, δράσει ενθαρρυντικά προκειμένου να υπάρξει πρόοδος ε, σχετικά με όλα αυτά τα θέματα χώρες όπως το Βιετνάμ είναι αναπτυσσόμενες, κινούνται προς τη ε, σωστή κατεύθυνση, αλλά ο δρόμος είναι δύσκολος. Ξέρουμε τι συμβαίνει με τις χώρες που ασκούν ε, υπερβολικά προστατευτικά ε, μέτρα. Και μια τέτοια συμφωνία θα ε, είναι θετική και για μας, όχι μόνο για το Βιετνάμ. Ο κύριος Σούστερ. Θεωρώ πως ε, μία κύρωση τη δεδομένη στιγμή δεν ε, είναι τη πράξη, διότι η πρόοδος όσο και ε, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, τόσο και στα, δικαιώματα, τα σταθερόμενα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που έχει να λάβει το κράτος δεν είναι παρκής. Χρειάζεται πολύ ε, χρόνος και πέρασε πολύς χρόνος από τότε που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις αλλά νομίζω πω ε, δεν έχουν γίνει τα βήματα με την ταχύτητα που θα έπρεπε να γίνει. Όλοι είδαμε πόσο χρόνο χρειάστηκε έτσι ώστε να υπογραφούν βασικές ε, συμφωνίε για, τα, ε, για βασικά πράγματα. Δυστυχώ η εμπειρία μας δείχνει ότι μέχρι, την, ε, μέχρι να έρθει η στιγμή της ακύρωσης θα περάσει πολύ καιρό και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να δίνει πρόσθετε ελαφρύνσει σε τρίτα κράτη τα οποία δεν σέβονται βασικέ διεθνεί συμβάσει. Δεν μπορούμε να λέμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ένα εμπόριο βασισμένο σε αξίες και στο τέλος ε, να αποδεικνύεται στην πράξη ότι το μόνο που ενδιαφέρει είναι η business. Δεν λέω βέβαια να διακόψουμε τελείω τι εμπορικέ μα σχέσει με το Βιετνάμ, αλλά όχι και να δώσουμε πρόσθετε ελαφρύνσει. Χρειάζεται πριν δοθούν αυτές οι ελαφρύνσεις ε, να υπάρχουν και διασφαλίσεις, ε, να υπάρξει και απτή βελτίωση. Να δούμε πρόοδο ουσιαστική. Γι' αυτό για μένα θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για την κύριο τη Συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σίγουρα δεν είναι και οι καλύτερε οι συνθήκε στο Βιετνάμ, αλλά πρέπει να βελτιωθούν. Εγώ έχω την αντίθετη άποψη ε, με το, από τον συνάδελφο. Αν δούμε τι γίνεται στα, με τα δικαιώματα των ε, γυναικών, θα δούμε ότι και εκεί υπάρχουν ε, προβλήματα. Το εμπόριο δεν μπορεί να λύσει βέβαια όλα τα προβλήματα. Χρειάζεται όμω να δημιουργηθεί μία βάση, μία αφετηρία. Δεν ξέρω πόσο φιλόδοξο είναι το Βιετνάμ, όμως ε, είχε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να καταφέρει να κάνει ουσιαστικά βήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι επιτέλους να σημειωθεί πρόοδος ε, ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα εργασιακά δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να πετήσουμε περισσότερα από την πλευρά του Βιετνάμ για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και θα μπορούσαμε να ασκήσουμε μέσω αυτής της συμφωνίας πίεση στο Βιετνάμ. Πιστεύω ότι το Βιετνάμ έχει δείξει ειλικρινές ενδιαφέρον για την βελτίωση των συνθήκων στους τομείς αυτούς. Θεωρώ πως ναι, πρέπει να παραμείνουμε σε ανοιχτό διάλογο, όμως να περιμένουμε με την κύρωση, διότι αυτά που συμβαίνουν ε, δεν είναι καλά. Δεν ε, πληρεί τις ε, προϋποθέσεις έτσι ώστε να να μπορέσουμε να κυρώσουμε την συμφωνία. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε με μεγάλη προσοχή την πρόοδο που σημειώνει το Βιετνάμ και μετά να πράξουμε. Jude και Darling έχει το λόγο. Θα συνεχίσω τα όσα είπε ο Γιώαχιμ και η Κάρολιν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ συγκεκριμένα και σαφή ορόσημο και μέτρα αξιολόγηση. Δεν με έπεισε η ακρόαση που έγινε στην Επιτροπή πριν από λίγο καιρό, όταν είχε έρθει ο υπουργό του Βιετνάμ και μας είπε ότι δεν υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στην υπογραφή της συμφωνίας και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει όμως ε, σχέση ανάμεσα στην υπογραφή της συμφωνίας και στην προστασία του περιβάλλοντος και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό προστίθεται σε όλες αυτές τις ε, αναφορές που έρχονται από πολύ αξιόπιστους διεθνείς οργανισμούς ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις αυξημένες πιέσεις κατά των ακτιβιστών στο Βιετνάμ. Θέλουμε να δούμε ένδειξη καλής θέλησης. Έχουμε δει ότι υπάρχουν και προβλήματα ε, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα του συνέρχεστε, στην ε, αναξιθρησκεία, η Διεθνής Αμνηστή αλλά και άλλες μη οργανώσεις έχουν αναφερθεί σε αυτό και τον περασμένο μήνα είχαμε και ένα καταπήγον ψήφισμα, το οποίο προψηφίστηκε μεγάλη πλειοψηφία στην ε, Ολομέλεια για, τα, για την κατάσταση των ε, δικαιωμάτων ακτιβιστών στο Βιετνάμ, μάλιστα. Και τότε είχαν πει οι συνάδελφοι ότι η κατάσταση είναι σαφέστατη. Ανθρώπινα δικαιώματα, σαφείς διατάξεις, άμεσα συσχετισμένες με την προστασία των επενδυτών και με την σχετική συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν τον Νοέμβριο έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως ήθελε να δει πρώτα πράξεις πρωτού προβεί σε κύρωση των συμφωνιών αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σαφήνεια τι προτίθεται να κάνει έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου και στο ψήφισμα που ενέκρινε τον Νοέμβριο και τι προτίθεται να κάνει σχετικά με όσα ακούσαμε για τη σύμβαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, για ε, το περιβάλλον και το πώς αντιδρά το Βιετνάμ σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σχολιάσει κάποιος. Κύριε Πρέσβη, θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα, το Βιετνάμ όσον αφορά την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Γι' αυτό θα ήθελα να ε, υπογραμμίσω ότι ουδέποτε στα Ηνωμένα Έθνη δεν έχει καταδειχθεί ε, το Βιετνάμ ε, ως μέρος της χώρας όπου γίνονται κατάφορες ή συστηματικές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων τα Ηνωμένα Έθνη ουδέποτε ενέκριναν συγγνώμη, ψήφισμα καταδικάζον το ε, ε, Βιετνάμ όσον αφορά τα προαναφερθέντα. Αναγνωρίζω ότι δεν είναι εξαιρετική η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο υπάρχουν και χώρες εντό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως όπου η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί Τέλεια. όσον αφορά τον εργασιακό κώδικα και τις συνθήκες εργασίας, υπάρχει ένας εργασιακός κώδικας στο Βιετνάμ, ο οποίος ε, τελεί υποσυζήτηση ε, στο Κοινοβούλιο του Βιετνάμ και η εκπόνηση του κειμένου ε, γίνεται σε στενή συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Όσον δε αφορά τις ε, θεμελιώδεις ε, συμβάσεις της Οργάνωσης Εργασίας, να σας πω ότι το Βιετνάμ συμμετέχει σε πέντε από τις πέντε παγκόσμιες συνθήκες για την οργάνωση εργασία. Υπάρχουν τρεις ακόμα συνθήκες για τις οποίες έχει εκδώσει η κυβέρνησή μου ήδη δικό χάρτη ε, εν ώψη της ένταξης της χώρας ε, και σε αυτές τις συμβάσεις. Ε, οι συλλογικές ε, συμβάσεις λοιπόν θα αποτελέσουν τον Οκτώβριο του 19 αντικείμενο ε, ψηφοφορίας ε, ε, από την Βουλή όσον αφορά την καταναγκαστική εργασία, όσον αφορά επίσης την ελευθερία επιλογής που επίσης θα τεθεί προέγκριση τον Οκτώβριο του 20 όσον αφορά τους μηχανικούς ε, διαλόγους ε, για το ανθρώπινα δικαιώματα. Γνωρίζετε, ε, φαντάζομαι, ότι το Βιετνάμ έχει ήδη υπογράψει μηχανισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στην ε, εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνεται μηχανισμός διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο διάλογος λαμβάνει η χώρα είτε στις Βρυξέλλες είτε στο Ανόη. Φέτος ο διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες και η βιετναμέζικη αντιπροσωπεία είναι και θα είναι στην διάθεσή σας στα πλαίσια του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων να ε, συζητήσει και με τους Ευρωπαίους βουλευτές για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μηχανισμός ε, εφαρμογής του ETCA που μελετάται στα πλαίσια της ε, ε, κοινής επιτροπής υλοποίησης της συμφωνίας και εντός αυτού υπάρχει η ειδική ομάδα η οποία ασχολείται με το κράτος δικαίου, τον, την καλή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η συγκεκριμένη υποεπιτροπή έχει αναλάβει την εκπόνηση τεχνικών προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βιετνάμ. Ε, όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν ότι ιδιαίτερος ενδιαφέρεται το Βιετνάμ ε, για τον διάλογο για θέματα ε, θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Peter Bertz from the Commission. Ευχαριστώ πολύ Peter από την Κομισιόν. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που βάλατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της ε, σημερινής σας συνεδρίας. Ευχαριστώ τους προλαλήσαντες, τον εισηγητή, την έκθεση. Ευχαριστώ για την έκθεση, ευχαριστώ για τις προτάσεις. Πολλά έχουν ε, υποθεί και δεν θέλω ε, να επαναλάβω τα ίδια. Να σας πω ότι ξεκίνησε η διαδικασία το 2012 ε, στα πλαίσια διαπραγματεύσεων με τις χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας, χώρες ΑΣΕΑΝ ε, και μετά από το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων με τη Σιγκαπούρη και την Μαλαισία. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε πάντα στενό ε, συνεργάτη του ε, Βιετνάμ και από τη δεκαετία του 90 όπου η ευρωπαϊκή κοινότητα είχε ξεκινήσει διαδικασίες συνεργασίας με την χώρα αυτή. Τρεις, τρία χρόνια πριν άρχισε να άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για την συμφωνία αυτή τη στιγμή η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών θα μπορέσει να αποτελέσει πλατφόρμα για περαιτέρω ανάπτυξη των επενδύσεων και του εμπορίου. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ευρύτερες γενικότερες σκέψεις ε, πριν σας δώσω μια μικρή σύνοψη του EVFTA. E-, e-, Οπωσδήποτε η συμφωνία, δεν χρειάζεται καν να το πω, ότι ενδυναμώνει τη σχέση μας εις την ε, Ασία, ε, όπου έχουμε ήδη ε, συμφωνίες με την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και την Κορέα. Η Κορέα είναι η μόνη η οποία λειτουργεί ήδη. Και ε, ε, πρόκειται για μια πρώτη συμφωνία περιφέρεια προς περιφέρεια Ευρωπαϊκή Ένωση με ε, και αποτελούν πρόδρομο για άλλες διαπραγματεύσεις με άλλες μεγάλες οικονομίες και χώρες ΑΣΕΑΝ. Επομένως, πρόκειται για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που οπωσδήποτε θα βοηθήσει ε, τις, ε, και τις χώρες οι οποίες έχουν ήδη ε, κάνει συμφωνίες με την ε, με χώρες ΑΣΕΑΝ, την Ινδία, την Κορέα, ε, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και οπωσδήποτε ε, στο τέλος αυτού του έτους στη συνολική και προοδευτική εταιρική σχέση του ειρηνικού. CPTPP. Όπως ε, είπαμε και προηγουμένως, αυτή η Συμφορία Ελεύθερων Συναλλαγών είναι η πιο φιλόδοξη και πιο συμπεριληπτική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αναπτυσσόμενη χώρα και αποτελεί ένα νέο μοντέλο ε, σχέσεων με την αναδυόμενη οικονομία. Θα ήθελα να πω ότι αυτό ισχύει και όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και όσον αφορά τα εργαλεία αλλά και όσον αφορά τις αξίες. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ε, προ... περιλαμβάνει και στοιχεία όπως ε, οι ελευθερίες, οι αξίες ε, και στοιχεία τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί στη συμφωνία με την Ιαπωνία. Βεβαίως γίνεται λόγος και για δασμούς και το Βιετνάμ θα αναιρέσει πολλές, πολλούς από τους υφιστάμενους εξαγωγικούς δασμούς ε, και ε, μέσω της ε, συμφωνίας θα διευκολυνθούν οι επαφές. Το Βιετνάμ επίσης θα ανοίξει στις ευρωπαϊκές εταιρείες την αγορά δημοσίων, τις δημόσιες, την αγορά δημοσίων συμβάσεων και θα διευρύνει επίσης τον τομέα των ε, υπηρεσιών. Η Κομισιόν έχει καταβάλει προσπάθειες να παρουσιάσει την ε, συμφωνία στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις ε, και αναγκαστήκαμε να τις χωρίσουμε σε δύο συμφωνίες. Τώρα όμως βρίσκονται οι συμφωνίες ε, στο τραπέζι. Η Κομισιόν ενέκρινε τη 17η Οκτωβρίου την συμφωνία και ε, στα αγγλικά και στις 12 Νοεμβρίου μεταφέρθηκαν και άλλες γλωσσικές εκδοχές ε, και δόθηκαν στο Συμβούλιο. Η συμφωνία ακολουθεί την ίδια αρχιτεκτονική και διάρθρωση με τη Συμφωνία της Σιγκαπούρης και παρομοίως με την Συμφωνία της ε, ε, Σιγκαπούρης είναι stand-alone agreement. Αλλά ε, βεβαίως χρειάζεται επικύρωση και ταυτόχρονη αποδοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συμφωνίες αυτές, όπως έχουμε πει ε, επανειλημμένα, ε, πρέπει να προχωρούν παράλληλα στα διάφορα θεσμικά όργανα ε, και επομένως οι νομικές υπηρεσίες της Κομισιόν ταυτόχρονα και παράλληλα με τις νομικές υπηρεσίες των χωρών μελών ελέγχουν την συμφωνία. Ε, και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του ελέγχου θα προχωρήσει ε, και η ΣΕΖΗΝ από πλευράς ε, του ε, Συμβουλίου. Να κάνω και μερικέ σκέψεις. Όταν έχουμε να κάνουμε με αναπτυσσόμενε χώρες όπως το Βιετνάμ, ε, ε, κανεί έχει δύο δρόμους, τον αποκλεισμό από τη μία και την συνεργασία από την άλλη. Είναι γεγονό ότι εμείς θέλουμε ένα ισχυρό Βιετνάμ, το οποίο όμως θα σέβεται το κράτος δικαίου. Ο, είναι γεγονός ότι εμείς ε, διαπιστώνουμε συγκεκριμένα στοιχεία ε, προόδου. Ε, είναι γεγονός ότι θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν μονάχα με αναφορές και εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιλέξαμε την ολιστική προσέγγιση. Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο ε, της ε, συμφωνίας ε, και έχουν πάντα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο όλων των εταιρικών σχέσεων και συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, διότι το κράτος δικαίου αποτελεί κύριο στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι και ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλωστε. Τις τελευταίες δεκαετίες υποστηρίξαμε το, στο Βιετνάμ πολλά προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ε, και για την πρόσβαση όλων στην δικαιοσύνη. Υπάρχει βεβαίως και ένα ε, κεφάλαιο που αφορά συγκεκριμένα επιπλέον μηχανισμούς ε, για περαιτέρω δέσμευση με το Βιετνάμ, έτσι ώστε ένα επιπλέον εργαλείο να μας δώσει την δυνατότητα συγκεκριμένης πρόοδου όσον αφορά τα θέματα αυτά. Τέλος, όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε ένα πολύ ισχυρό ε, κεφάλαιο TST και είμαστε πεπισμένοι ότι δεν είναι δυνατόν ε, να έχουμε οικονομική ανάπτυξη ε, που όμως θα ζημιώνει το περιβάλλον ή τα εργασιακά. Και γι' αυτό ζητούμε την συμφωνία του Βιετνάμ όσον αφορά τις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου, Εργασία, Εργασίας. Συγγνώμη. Όπως είπε και ο πρέσβης ε, προηγουμένως, ε, γίνεται προσπάθεια, ε, μια προσπάθεια την οποία επιτείνει και η Επίτροπος Μάλστρομ στις επαφές που έχει ε, με, με τον πρέσβη και τους λοιπούς αξιωματούχους του Βιετνάμ. Ευελπιστούμε επομένως ότι και το Βιετνάμ θα ξανασκεφτεί όλες τις δεσμεύσεις που πρέπει να έχει στην εθνική του νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα μεταφέρω όλα αυτά στον ε, κύριο Ζαραντέλε, κύριο Κάμπελε. Νομίζω ότι θα πρέπει με, με δικαιοσύνη ε, να αντιμετωπίσουμε ε, το Βιετνάμ και να δούμε συνολικά το ζήτημα, έστω και αν έχουμε κάποιες ε, αντιρρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τα έχουμε όλα λοιπόν τώρα στο τραπέζι λέει ο Πρόεδρος. Είναι συγκεκριμένο το αίτημα του Κοινοβουλίου προς την κυβέρνηση ε, του Βιετνάμ και περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένες ε, δεσμεύσεις. Φτάνουμε λοιπόν στην προθεσμία Υποβολή τροπολογιών 15 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα. Έχετε αρκετό χρόνο ε, και στις ε, χριστουγεννιάτικες ε, διακοπές να τα σκεφτείτε όλα αυτά. 6 το απόγευμα στις 15 Ιανουαρίου. Επόμενο θέμα, προστασία επενδύσεων του Βιετνάμ. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό ε, το έχουμε αντιμετωπίσει. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος ε, συνάδελφος να ξαναπάρει το λόγο συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Όχι από ό,τι βλέπω. Και επομένως να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση αυτή. ίδια ε, η ίδια προθεσμία 3η 15 Ιανουαρίου και ε, για την προστασία των επενδύσεων. Πάρα πολύ ωραία άψογα. Επόμενο θέμα είναι τα διάφορα. Ξέρετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα ξέρετε όλα αυτά. Είναι αυτό το δέντρο στο ισόγειο και έχουμε και μία έκτακτη συνεδρίαση την 10η Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Γιατί έχουμε μερικά πολύ σημαντικά θέματα να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.